Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ να καθίσετε και θα ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Your motion for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 Uh, Ας ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίσεώς μας. Είναι ε, μία ασυνήθιστη ιστορική στιγμή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε μια κοινή επιτροπή της ευρείας εκπροσώπησης των κρατών μελών, δηλαδή των Υπουργών Γεωργίας, της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συζητήσουμε την κοινή αγροτική μας, γεωργική μας πολιτική, μία από τις πλέον παλές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω καταρχήν τον Υπουργό κύριο Σαβίσκη ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωργίας και τον κύριο Τσόλος που είναι ο Επίτροπος Γεωργίας και όλους εσάς που είσαστε εδώ Υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών. Ε, είμαστε σε κοινή συνεδρίαση με τον συνάδελφο πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κυρίου Κάστρο και χάρη στον κύριο Σαβίσκη και τον κύριο Ντεκάστρο έχουμε αυτό το ασυνήθιστο γεγονός και θέλω να συγχαρώ όλους τους παρόντες. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό επίτευγμα, μάλλον στα σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, ε, ο καθένας δε από εσά μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα, διότι και εγώ το ίδιο ετοιμάζομαι να κάνω. Κυρίες και κύριοι, και πάλι θα ήθελα να σας καλωσορίσω διότι θα επεξεργαστούμε την ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ε, ε, αναμόρφωση της κοινή γεωργικής πολιτικής που είναι από τις παλαιότερες πολιτικές μας. Θέλω να ε, συγχαρώ την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που συνέταξα τον Ιούνιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία νέα πρόταση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής για την προσαρμογή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και εφαρμόζοντας τις, τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα έχει ισχυρά αγροκτήματα τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά και θα έχει και μια ισχυρή γεωργία εφόσον η γεωργία είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να εξέλθουμε αυτή της κρίσεως γρήγορα. Η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει ιδιαίτερα προνόμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη γεωργία, με τις δημοσιονομικές αποφάσεις, και τις αποφάσεις που άπτονται της γεωργίας και της αλίας. Έχουμε λοιπόν συνενώσει τις δυνάμεις μας κατά τρόπον ώστε να λαμβάνουμε κοινέ αποφάσεις και συγχρόνως οι συζητήσεις αυτές και οι αποφάσεις να είναι διάφανες, να γνωστοποιούνται και να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό, να είμαστε σε στενή επαφή με τους πολίτες, να καταλήγουμε από κοινού στις ευρωπαϊκές αποφάσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια Ευρωπαίων και αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Θέλουμε η γεωργία μας να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική και να την καταλήγουμε καταστήσουμε πιο ε, στραμμένη ε, προς την κοινότητα και ε, ιδίως να συντονίσουμε τις μικρές και μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης με αυτές που είναι στην περιφέρεια, αυτές που είναι στο βορρά, με αυτές που είναι στο νότο. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκμετάλλευσης, διαφορετικές εξελίξεις και θέλουμε κοινή γεωργική μας πολιτική να λάβει υπόψη όλες τις πτυχές του περιβάλλοντας, ε, να προωθήσουμε τη γεωργική παραγωγή, να ζούμε μια υγιεινή ζωή και η ύπεθρος να μπορέσει να καταστεί ε, ευχάριστη για να ζει κανείς ευχαρίστως εκεί όπως και στις πόλεις. Άρα η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι πολύ σημαντική για μας και είμαι πεπισμένος ότι οι συζητήσεις τις οποίες ξεκινούμε τώρα με τόσο ευρύ τρόπο είναι απλώς μία συνέχιση του τι έχει γίνει εδώ και μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον και εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλές συνεδριάσεις, σε πολλά μέλη. συνήθως συνοδευόμενος από τον Επίτροπο Τσόλος και από άλλους εκπροσώπους των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να προετοιμάσουμε τη σημερινή συζήτηση και έχουμε μία βαθιά κατανόηση διαφόρων προβλημάτων και των λύσεων που μπορούμε να επιλέξουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τις καλύτερες ευκαιρίες στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απευθύνουμε σε εσά. Είσαστε ειδικοί. Εσείς θα αποφασίσετε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η ΚΑΠ και θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, να καταλήξετε σε καλές λύσεις, να έχετε επικοδομητικές συζητήσεις και να μας συνοδεύσουν στις αποφάσεις μας οι πολίτες που είναι κάτι πολύ βασικό για μας σήμερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κύριο Μπούζεκ για την τιμή που μας κάνει σήμερα να βρίσκεται εδώ και να κηρύξει την έναρξη εργασιών αυτής της έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας από κοινού με, του, με όλους τους Υπουργούς Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν ε, δείχνει πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή όπου όλοι καλούμεθα να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις ε, στο μέλλον των ε, Ευρωπαίων Γεωργών. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και σας καλωσορίζουμε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση για τη μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Για πρώτη φορά έχουμε εδώ κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας και της Επιτροπής για τη Γεωργία και την ε, ανάπτυξη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια συνάντηση που καταδεικνύει το ότι είναι ιδιαίτερη η σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. σε αντίθεση με το παρελθόν. Το, κατά το παρελθόν υπήρξε ένα κύκλο που ξεκίνησε το 1992 και ο οποίο βασιζόταν σε μια λογική τη συνέχεια, η οποία καθίστε το δυνατή από το γεγονό ότι για 50 ολόκληρα χρόνια είχαμε αποκλίνουσες τιμέ των πρώτων υλών τη γεωργία με τι τελικέ τιμέ. Σήμερα όμω τα πράγματα έχουν τελείω αλλάξει. Η Ευρωπαίοι γεωργοί όπω και υπόλοιποι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς καταστάσεις γιατί και στις ανεπτυγμένες περιοχές ε, έρχεται, επανέρχεται ο εφιάλτης της ε, έλλειψης τροφίμων. Οι αγορές χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις, ε, οι οποίες ε, στο μέλλον ενδέχεται να εξελιχθούν και σε συστηματικές. Το δικό μας το σύστημα της ε, προσφοράς θα δοκιμαστεί σκληρά κατά τα επόμενα έτη και οι φιλοδοξίες των πολιτών και όσων χαράσουν πολιτική, οι φιλοδοξίες αυτές σχετικά με τη γεωργική πολιτική βρίσκονται και αυτές υπό μεγάλη δοκιμασία. Εμείς επιθυμούμε να έχουμε μια γεωργία η οποία θα διασφαλίσει συνέχεια του εφοδιασμού, παράλληλα όμω θα σέβεται τα βασικά αγαθά όπω είναι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, η ε, πολιτική φιλική προ το περιβάλλον, η κοινωνική συνοχή. Πεθυμούμε πάνω απ' όλα μια οικονομία, μια γεωργία η οποία θα είναι βιώσιμη ε, με βάση οικονομικά κριτήρια. Αυτό που σήμερα είναι η ευθύνη μα είναι πάνω απ' όλα να προσφέρουμε στον γεωργικό τομέα και στους γεωργού μα τα εργαλεία εκείνα που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση που είναι να παράγουν περισσότερο με λιγότερη μόλυνση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί και περαιτέρω γεωργικό δυναμικό. Είναι λοιπόν καθήκον μας να χαράξουμε τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίοι θα επιτρέπουν στους γεωργούς μας να είναι πιο ισχυροί, πιο ανταγωνιστικοί, να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τα νέα σενάρια αστάθειας των αγορών, οι οποίες αγορές συμπιέζουν το εισόδημα των γεωργών και μάλιστα πολλές φορές απειλούν ακόμα και την επιβίασή τους. Οι προτάσεις που πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκάλεσαν έντονη κριτική τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο επικρατεί μία σύγχυση. Όσον αφορά τις προθέσεις της Επιτροπής Επικοινωνίας στις 18 Νοεμβρίου του 2008, κάτι το οποίο το εκτιμήσαμε βέβαια, εμείς δεν θεωρούμε ότι οι προτάσεις αυτές είναι τόσο φιλόδοξες όσο θα έπρεπε να είναι. Κατά τις πρώτες συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην Επιτροπή Γεωργίας, τη δική μας, κατέστη απόλυτα σαφές ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις συνθήκες που έχουν αλλάξει. Και δεν πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Τα μέτρα που προτείνονται μοιάζουν όμως να ακολουθούν τη συγκράτηση της παραγωγής και όχι την αύξησή της. Το γραφειοκρατικό άχθος για τους γεωργούς, τουλάχιστον κατά την άποψη των περισσότερων πολιτικών ομάδων, να εντείνεται περαιτέρω. Τα μέτρα λοιπόν για να αντιμετωπιστούν, ε, αντιμετωπιστεί η κρίση, τα μέτρα αυτά μοιάζουν ανεπαρκή. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε χαράξει ένα φιλόδοξο δρόμο. Ε, το δρόμο αυτό τον χαράξαμε με δύο εκθέσεις, η μία ε, του Ευρωβουλευτού Λιών και η άλλη του κυρίου Ντες, έχοντας ως στόχο να σεβαστούμε την εντολή που μας έδωσε η ευρύτατη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, η οποία ενέκρινε αυτές τις δύο εκθέσεις. Όμως και οι Ευρωπαίοι πολίτες μας έχουν δώσει και αυτή μια εντολή μέσα από την συναπόφαση. Και με αυτήν την συναπόφαση είμαστε πλέον υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την νομοθετική διαδικασία. Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε σήμερα ακολουθεί μια κατεύθυνση διαφανή, κοινή και ελπίζω αυτά να μην είναι τυχαία. Η συζήτηση θα μας βοηθήσει να αναζητήσουμε από κοινού τη σύγκληση για να ξεπεράσουμε τα όρια της πρότασης που έχει κατατεθεί και να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε. Ζητάμε από την Επιτροπή να μας συνδράμει σε αυτό μας το καθήκον και να επιταχύνει τη συμφωνία. Ελπίζουμε να συναυτεί αυτή σύντομα. Ε, θέλω να σας πω και νομίζω εδώ έχω και την ε, σύμφωνη γνώμη της ε, πλειοψηφίας της Επιτροπής ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα απεκδηθεί των ευθυνών του και δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των προνομίων του οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο και οποτεδήποτε κρίνουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Ευχαριστώ όλους σας και θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας βεβαίως τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σαβίκη, για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει, για τον διάλογο που ε, ακολούθησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και βεβαίως ευχαριστώ και όλους τους ε, παριστάμενους υπουργού Γεωργίας και τον Επίτροπο κύριο Τσόλος, ο οποίος όπως ε, πάντα είναι διαθέσιμος για τον διάλογο που πολλές φορές είναι και αρκετά έντονος ο διάλογος αυτός. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου ευχαριστώντας τους εισηγητές στους οποίους ε, το Κοινοβούλιο ανέθεσε να συντάξουν την έκθεσή του. Τον κύριο Καπούλα Σάντος από τους Σοσιαλιστές και τον Μισελ Νταντέν και τον Τζοβάνι Λαβία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Σαβίτσκι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτοί οι υπουργοί, αξιότιμοι προσκαλεσμένοι, όλα καλά, ωραία. Κύριε Πρόεδρε. Βυσόκα Κομίσιο, και Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπούζεκ, είπατε μόλις πριν από λίγο ότι αυτή η συζήτηση έχει ιστορική σημασία. Αυτό είναι αληθές για τρεις λόγους. Εμείς ως Προεδρία εφαρμόζουμε τους κανόνες που απορρέουν από τη Συνδίκη της Αβώνας σε ό,τι αφορά την ε, συναπόφαση. Ε, ξεκινάμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και τρίτον είναι η πρώτη πολωνική προεδρία από τότε που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τρεις λόγους λοιπόν είναι ιστορική σημασία σε αυτή η συζήτηση. Η ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου στη Βαρσοβία το Σεπτέμβρη Ε, την ε, πρωτοβουλία ανέλαβε ο κύριος Ντεκάστρο, πρόεδρος, και ο Επίτροπος Τσιόλος και βέβαια ε, ο ίδιος ο υποφαινόμενος, οι τρεις μας μαζί. Αποφασίσαμε τελικά να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής η οποία είναι όλο και πιο περίπλοκη, και όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί, διότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος και του παρόντος, να ικανοποιήσει τις επιθυμίες όλων των εμπλεκομένων και να συνδυάσει τα συμφέροντα ε, και των παραγωγών και των γεωργών. Ε, αποφασίσαμε αυτός, αυτή η συζήτηση να γίνει σε τρεις ημερομηνίε. Η πρώτη μεταξύ ευρωβουλευτών και Υπουργών Γεωργίας οι ε, ε, επόμενοι με συναντήσεις των ε, γεωργών, των, των κατεξοχήν ενδιαφερομένων δηλαδή, και την ε, Κεμιτρίτη τρίτη θα λάβει χώρα ε, με τους εμπειρογνώμονες. Οι επόμενες δύο στις 23 Ενδεκάτου και στις 7 Δωδεκάτου. Σήμερα 23 Ενδεκάτου και 7 Δωδεκάτου. Η πρώτη παρουσίαση του νομοθετικού πακέτου 7 κανονισμών έγινε από τον κύριο Τσιόλος τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών τότε έγινε και μια πρώτη προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε, έγιναν οι προτάσεις ε, δεκτές ε, με πολύ ενθουσιασμό από τους υπουργού. Τώρα περνάμε σε ένα επόμενο επίπεδο πλέον συζήτηση των προτάσεων. Σε μια εβδομάδα, όταν ξανασυνέλθει το Συμβούλιο, θα συζητήσουμε το θέμα σε βάθος, θα συζητήσουμε το θέμα των άμεσων πληρωμών επίσης το Δεκέμβρη και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Αυτή, αυτό είναι και το χρονοδιάγραμμα που έχει προτείνει η Πολωνική Προεδρία. Ο δρόμος ε, είναι δύσβατος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ έτσι ώστε να επιτύχουμε μια σύγκληση απόψεων. Είναι προφανές ότι η πρόκληση, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, έχουμε περιβαλλοντικές προκλήσεις, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό δυσκολιών και πολύ ψηλές προσδοκίες να αντιμετωπίσουμε. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε τους ε, κανόνες της ε, συνθήκης, τους οποίους θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε απαραίτητα. Η πρόταση της ε, Κομισιόν αποτελεί σημείο εκκίνησης. Όλοι μαζί θα πρέπει να καθορίσουμε την καινούργια κοινή αγροτική πολιτική ε, ένα θέμα το οποίο η Πολωνική Προεδρία το έχει οθετήσει ως βασικό θέμα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της. Θα πρέπει η καινούργια ΚΑΠ να είναι πιο απλουστευμένη και να προσαρμόζεται καλύτερα στις ε, μελλοντικές προκλήσεις. Θα πρέπει να καθιστά την Ευρωπαϊκή Γεωργία πιο, αποτελε... πιο ε, ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή και βιώσιμη. Ευχαριστώ πολύ που διαργανώσατε τη σημερινή συνάντηση. Αυτή την αρχή του διαλόγου είναι μια, μια πολύ ε, καλή και θετική κίνηση. Ελπίζω ότι θα οδηγηθούμε σε μια πραγματικά καλύτερη ΚΑΠ. Ε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που οργάνωσαν αυτή τη συζήτηση μετά από την υποβολή των προτάσεων για την αναθεώρηση της ε, γεωργικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ τον πρόεδρο Μπούζεκ για την, πολιτική, για την προσοχή που αποδίδει σε αυτή την πολιτική η οποία είναι η μόνη πραγματικά κοινοτική με οικονομικό χαρακτήρα και είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως σε αυτή τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως άρα το να δοθεί η δυνατότητα συζητήσεως μεταξύ του Συμβουλίου και και ε, ε, του, Συμβουλίου, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου θα ε, εφαρμόζει και προωθεί την συναπόφαση για μια κοινοτική πολιτική η οποία θα είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη τομεακή πολιτική γιατί ό,τι αποφασίσουμε από κοινού θα εφαρμοστεί σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε περιοχή. Εξού και χαίρομαι που βλέπω πόσο ζωντανή είναι η συζήτηση στο θέμα αυτό. Βρίσκω ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία ζωντανή συζήτηση. Ξεκίνησε η δημόσια συζήτηση στο τέλος του χρόνου πέρυσι και το τώρα προωθούμε τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι και θα πρέπει να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Δηλαδή όχι μόνο να αποφασίσουμε επί ενός ή άλλου σημείου αλλά επί το συνόλου. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική. Δεν μπορεί να επιλέξουμε μόνο ό,τι μας αρέσει και να αφήσουμε ό,τι δεν μας αρέσει. Θα πρέπει εφόλης της ύλη να υπάρξει μία απόφαση, μία συνεκτική πρόταση για να παραμείνει συνεκτική και η ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι θα ληφθούν πολιτικές αποφάσεις αλλά βάσει τεχνικών μέσων τα οποία θα εφαρμοστούν επιτόπου. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα με πολλές σελίδες, πολλά στοιχεία και είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών διότι λαμβάνουμε πολιτικές σχέσεις στο ένα σημείο ή στο άλλο αλλά θα πρέπει καταρχήν να αντιληφθούμε τι έχει προταθεί. Γι' αυτό και όλες οι συζητήσεις αυτές, όλα αυτά ε, τα συνέδρια που έχουν ε, προτείνει ο Πάολο Ντεκάστρο και ο κύριος Σαβίσκι για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ χρήσιμα καθότι θα μας επιτρέψουν να αναλύσουμε τις προτάσεις αυτές και να κατανοήσουμε τι υπάρχει προσυζήτηση. Ε, άκουσα πολλές αντιδράσεις που είναι φυσιολογικές. Ο καθένας εκφράζεται γιατί θα εμπλακεί στη λήψη αποφάσεων και πολλές φορές είδα στον θέματα να συζητούνται που δεν έχουν ακόμη αναλυθεί και παρατηρήσεις για προτάσεις που δεν έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή συμπεράσματα για στοιχεία που ποτέ δεν παρουσιάστηκαν έτσι στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξού και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε περαιτέρω στο πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι συνεκτικό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω κύριε Ντεκάστρο ότι αυτό που υπάρχει στο τραπέζι, αυτό που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλήρως συνεκτικό με ό,τι περιείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση πέρυσι τον Νοέμβριο. Μπορεί να μην συμφωνούμε με ορισμένα στοιχεία αυτής της πρότασης, αλλά λαμβάνουμε υπόψη το θέμα της ε, παραγωγής τροφίμων θέλουμε να υποκινήσουμε τους γεωργούς να αυξήσουν βιώσιμα την παραγωγή με ε, άμεσες ενισχύσεις στα εισοδήματα και κίνητρα για να υπάρξει μία βιώσιμη αύξηση της παραγωγής μέσω των γεωργών, διότι αποτελούν όλα τα μέτρα αυτά μια συνολική θεώρηση η οποία περιλαμβάνει και τις ανάγκες των γεωργών για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, αλλά πάντα και στις προσμονές των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι η κοινή η γεωργική πολιτική η οποία είναι δημοσία και αν δεν μπορέσει να συγκεράσει τα δύο συμβαλόμενα μέλη δηλαδή αφενός τους γεωργούς οι οποίοι θα χαίρουν άμεσα αυτή τη ενίσχυση και τους καταναλωτές που θα χαίρουν τη στηρίξεως με την βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου εάν δεν ικανοποιήσουμε και τις δύο πλευρές απλώς θα ενισχύσουμε τις ε, διαφορές που υπάρχουν και τα κενά που υπάρχουν αφενός μεταξύ των γεωργών και αφετέρου μεταξύ της κοινωνίας της Ευρώπης. Και δεν έχουμε δικαίωμα να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να υπεραμεινθούμε των γεωργών για να κάνουν το καθήκον τους στην Ευρώπη και αυτή είναι και η έννοια της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σύντομα θα επανέλθω στο θέμα αυτό της ισορροπίας μεταξύ μεγαλύτερης παραγωγής και βιώσιμης χρήσεως των πόρων, διότι όπως είπατε ακούσαμε ότι η μελλοντική ΚΑΠ θα εμπροδίσει την παραγωγή ενώ πρέπει να διπλασιάσουμε την παραγωγή στο μέλλον. Άλλοι λέγουν ότι με τα μέτρα του περιβάλλοντος που έχουμε προτείνει απλώς ε, κάνουμε ένα washing, ένα πράσινο ξέπλυμα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες ε, για πρώτες ύλες. Υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή και αυτό αποδεικνύει ότι κατά βάθο κάπου πρέπει να υπάρχει μια ισοσκελισμένη η οποία στηρίζει τη γεωργική παραγωγή και συγχρόνως ε, ενθαρρύνει τους γεωργούς να ακολουθήσουν μία βιώσιμη μέθοδο και από την άλλη πλευρά ο μόνος λόγος της πολιτικής να μην είναι η διαχείριση των τοπίων αλλά και της συλλογικής διαχειρίσεως των γεωργικών γεών με μία βιώσιμη προοπτική. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες προσπάθειες για να εφαρμόσουμε την έρευνα και την καινοτομία για να αυξήσουμε την γεωργική παραγωγικότητα. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και δεν έχουμε άλλη λύση στο μέλλον για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα κατά τρόπον βιώσιμο και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε επιτόπου τα αποτελέσματα των ερευνών. Πρέπει λοιπόν να διαπιστωθεί η προσπάθεια που έγινε για να εντοπίσουμε ένα σωστό προϋπολογισμό για τη διατροφή και τη γεωργία. Και τώρα εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλέον αποτελεσματική χρήση αυτού του προϋπολογισμού και να εξασφαλίσουμε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής θα γίνει αποτελεσματικά, ορθολογιστικά, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουμε σε επιστημονικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά διατηρούμε μία ιδιαίτερη στήριξη για τις μειονεκτικές περιοχές για να υπάρχει εκεί κάποια προώθηση και γι' αυτό τονίσαμε στην πρότασή μας τη στήριξη για τις μειονεκτικές περιοχές και αποφασίσαμε να διατηρήσουμε και να διατυπώσουμε καλύτερα το συνδυασμό των μέτρων όπου στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν οι παραγωγές ή παραγωγή λόγω των συνθήκων παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα μέτρα τίνουν στο να στηρίξουν την παραγωγή και να αυξήσουν την παραγωγή. Απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι έχουμε καταρτήσει μόνιμα μέσα για τη διαχείριση της αγοράς βάσει αυτών που έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Η ε, αγορά να αποτελέσει πραγματικά ένα δίχτυ ασφαλείας και θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Τώρα όμως θα σταθώ στην οικολογική ανταγωνιστικότητα του πρώτου πυλώνα και πιστεύω ότι είναι βασικό να εξετάσουμε τις επιδόσεις στο μέλλον και ε, στη γεωργία χωρίς όμως αυτό να είναι εις βάρος των πρώτων υλών και ε, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει αντίφαση με την χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων διότι το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αν το τομνήσουμε σαφώς με αρχές που βασίζονται στη δημόσια πολιτική η οποία ακολουθεί τη γεωργία βαίνουμε προς το συμφέρον των γεωργών διότι αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την παραγωγή Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, αλλά στην Ευρώπη δεν μπορεί να αυξήσει κανείς την παραγωγή αυξάνοντας τις εκτάσεις, αλλά βελτιώνοντας τις εκτάσεις τις οποίες εκμεταλλευόμαστε και καλλιεργούμε. Πρέπει να συνδέσουμε τα δύο αυτά στοιχεία και τα μέτρα που έχουμε προτείνει έχουν προταθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε αποτελέσματα χωρίς να αυξήσουμε υπερβολικά το διοικητικό φορτίο και εδώ αναφέρομαι στο διοικητικό άχθος το οποίο αυξάνεται διότι είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρόνως να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού σε κάθε πολιτική. Και είναι σωστό, για να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να καθορίσουμε σαφείς στόχους. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα δώσουμε χρήματα χωρίς να ζητάμε τίποτα εις αντάλλαγμα. Αλλά το Κοινοβούλιο, το οποίο φυσιολογικά είναι υπόλογο εις τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους για την διαχείριση ενίσχυση των ε, ευρωπαϊκών δημοσιονομικών μέσων ε, ζητά πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι για να υπάρξουν αποτελέσματα. Και όταν προτείνουμε ορισμένα μέτρα θέλουμε να υπάρξουν αποτελέσματα και αυτό να γίνει με το πλέον απλό και εύκολο τρόπο η απλοποίηση που αναφέρονται πάλι στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού άχθους. Εάν δείτε το πρόγραμμα της αναπτύξεως της υπαίθρου, έχουμε προτείνει νέα μέσα για να υπάρχει ευελιξία στα κράτη-μέλη και να μπορέσουν τα μέτρα αυτά να χρησιμοποιηθούν με το πιο απλό δυνατό τρόπο. Δηλαδή αυτό που φέρνουμε στο τραπέζι είναι μία εύκολη μέθοδος προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κρατών των μελών ε, ε, προσπαθώντας να απλοποιήσουμε. Είχαμε επίσης αναφερθεί τα διοικητικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την πολλαπλή συμμόρφωση και πρέπει να πούμε ότι στο σημείο αυτό τα κράτη και οι περιοχές οι οποίες χρησιμοποιούν σωστά τους πόρους θα μπορέσουν να μειώσουν και τους ελέγχους εάν γίνεται σωστή χρήση αυτών των διοικητικών μέσων και οικονομικών πόρων. Άρα βελτιώνουμε και τους ελέγχους. Υπάρχει το πρόγραμμα πληρωμών για τους μικρούς γεωργούς που απλοποιεί τους ελέγχους για 33% των αποδεκτών της ΠΑΚ αλλά καλύπτει μόνο ένα μικρότερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων και έτσι θα μειώσουμε το κόστος και για τις διοικήσεις αλλά και για τους γεωργούς. Και τέλος τα μέτρα τα οποία ε, έχουμε προσαρμόσει και προτείνει για το πρασίνισμα, αν θυμάστε είχαμε συζητήσει διάφορα θέματα όταν έγινε η δημόσια διαβούλευση και προτείναμε μόνο τα μέτρα που είναι εύκολο να ελεγχθούν. Και εδώ αν δούμε τους στόχους τους οποίους καθορίσαμε μέσω αυτών των μέτρων που προτείνουμε στην κοινή γεωργική πολιτική ε, και το διοικητικό άχθος θα διαπιστώσετε ότι δεν έχει αυξηθεί το κόστος αυτό ενώ θα μπορούμε να αποδείξουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι και ποια είναι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε μέσω αυτών. Τέλος, η διαχείριση των αγορών και με αυτό θα τελειώσω. Ήμασταν πιστοί σε αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει στις διάφορες συζητήσεις να ενισχύσουμε το μηχανισμό της αγοράς σαν δίχτυ ασφαλείας που μας επιτρέπει να προβλέψουμε τις κρίσεις, να επεμβαίνουμε στις της και με την ε, χρήση των ε, παραδοσιακών ε, μέτρων δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθήκευση συν έκτακτα μέτρα να μπορούμε να δράσουμε γρήγορα όταν υπάρχει μια κατάσταση κρίσεως. Συγχρόνως προτείνουμε μέτρα που δεν προϋπήρχαν και δεν υπάρχουν τώρα για να διαχειριστούμε δύο δύσκολες καταστάσεις στην αγορά. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με το βάρος που θα αποδώσουμε στις οργανώσεις παραγωγών για την καλή λειτουργία των αγορών, θα δείτε μία προώθηση στο μέλλον μια καλύτερης διαχείρισης των αγορών, όχι μέσω μεγαλύτερης ε, γραφειοκρατίας και διοικητικής πιέσεως και εμπλοκής της δημοσίας διοικήσεως αλλά με μεγαλύτερης εμπλοκής των ενδιαφερομένων στη σωστή διαχείριση της αγοράς και αν τους εξοπλίσουμε και με τα οικονομικά μέσα για να μπορέσουν να συνεργαστούν, νομίζω ότι θα υπάρξει και μία χρηστή διαχείριση των αγορών, αφήνοντας τις αγορές να δώσουν το σωστό μήνυμα προς τους παραγωγούς. Αυτά είναι ορισμένα στοιχεία τα οποία ενισχύουν την ιδέα ότι η πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ισοσχελισμένη, απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών, στην ε, ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας με στόχο να διατηρήσει τη συνεκτικότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Βεβαίως, Πάολο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι παρούσα για να προσφέρει κάθε βελτίωση της πρότασης, αλλά αυτό όμως τώρα ε, που ζητώ είναι να αναλύσουμε τις προτάσεις που είναι στο τραπέζι, είναι τεχνικές, αλλά ε, θα χρειαστεί πολιτικός διάλογος για να καταλήξουμε ε, σε μέτρα τεχνικά που θα εφαρμοστούν επί τόπου με τρόπο απλό και αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση. Non avremo Αγαπητέ Επίτροπε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την συνεργασία που θα έχουμε με την Επιτροπή και με τις ε, υπηρεσίες και με το, τους συνεργάτες για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στα διάφορα θέματα της Γεωργίας. Θα περάσουμε τώρα κανονικά θα έπρεπε να περάσουμε ε, στην Υπουργό Γεωργίας της Δανίας. Ε, δεν ήρθε όμως και κάποιο πρόβλημα με το αεροπλάνο. Θα δώσω το λόγο στον Κύπριο Υπουργό Γεωργίας. Παρακαλώ, έχει το λόγο ο κύριος Σοφοκλής Αλετράρης κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. καταρχή θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε τη σημερινή συνάντηση και να ευχαριστήσω ταυτόχρονα για την ευκαιρία που μου δίδεται να προσφωνήσω στη συντομία την Επιτροπή σας ως μέλος του Τρίου της παρούσας Προεδρίας του Συμβουλίου. Όλοι έχουμε επίγνωση της μεγάλης σημασίας που έχει η στενή συνεργασία μεταξύ των δύο σωμάτων μας για διασφάλιση της καλής λειτουργίας των θεσμών και για την πρόθεση και ολοκλήρωση της επιθύρας μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, της πιο ανεπτυγμένης και της πιο σημαντικής ίσως κοινή πολιτικής που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει προτάσεις που προδιαγράφουν μία πλούσια σε εύρος και σε λεπτομέρεια μεταρρυθμιστική προσπάθεια και θέλουμε την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Επίτροπο Τσιόλος για την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει ο ίδιος και οι υπηρεσίες του για την ετοιμασία τους. Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών είναι μεγάλες, οι προκλήσεις πολύπλοκες και οι καιροί δύσκολοι. Θα πρέπει όλοι να εργαστούμε με σύμπνοια και συναντήληψη για να φέρουμε σε αίσιο πέρα στο δύσκολο αυτό έργο. Η Κύπρος θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου στο δεύτερο εξάμεινο του 2012 και φιλοδοξεί με τη δική σας σύμπραξη και συμβολή και με τη συμπαράσταση των δύο άλλων μελών του Τρίου Προεδρίας, της Πολωνίας και της Δανίας, να ολοκληρώσει πριν το τέλος του 2012 τη συζήτηση και τη ψήφιση των βασικών κανονισμών που διέπουν την κοινή γεωργική πολιτική. Είμαστε μια μικρή χώρα με περιορισμένους πόρους και δυνατότητες και έχουμε επίγνωση της πολυπλοκότητας των θεμάτων που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Ταυτόχρονα όμως είμαστε και μια χώρα που δεν έχει μεγάλα συμφέροντα για να τα προωθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Προσβλέπουμε λοιπόν να συμβάλλουμε θετικά, ουδέτερα και επικοδομητικά στην εξυπηρέτηση των κοινών στόχων, αναλαμβάνοντας με πλήρη διαφάνεια και καλή θέληση το ρόλο του δίκαιου μεσολαβητή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια αυτά θέλω να τονίσω εξ αρχής και χωρίς να προκαταλαμβάνω την παραπέρα συζήτηση ότι ως Κύπρος αντιμετωπίζουμε θετικά τις βασικές προθέσεις και τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύγκληση και συμβολή στην κοινή στρατηγική του 2020, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη, δικαιότερη κατανομή των πόρων με βάση αντικειμενικά κριτήρια, μεγιστοποίηση της προσφοράς δημοσίων αγαθών και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων της ευρωπαϊκής γεωργίας και ενίσχυση των μικρών παραγωγών, συνεργασία και συντονισμός με τα διαρθρωτικά ταμεία για ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, αξιοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς χρειαζόμαστε τους ανάλογους πόρους και κατά συνέπεια η συζήτηση και αποτελεσματική διεκπαιρέωση των θεμάτων που σχετίζονται με το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο έχει για μας ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει όλοι από κοινού να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον παράλληλο αυτό τομέα και να μην θεωρούμε τις προτάσεις της Επιτροπής ως τελεσίδικες και δεδομένες. Επί του προκειμένου, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για το θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τη συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η κοινή γεωργική πολιτική για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020. Ταυτόχρονα θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι με τη στενή συνεργασία και τη συμβολή όλων των φορέων και θεσμών θα καταστεί δυνατόν όπως οι καλές προθέσεις και βασικές αρχές που διέπουν τις προτάσεις της Επιτροπής μεταφραστούν τελικά σε καλές, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις έχοντας σαν βασικό αξίωμα την απλοποίηση και τη μείωση του διοικητικού άκθους. Έχω γράψει, κύριε Τσόλο, τη λέξη απλοποίηση με κεφαλαία για να τονίσω ότι θα πρέπει να μην παραμείνει στη σφαίρα της θεωρητικής διακήρυξης. Το αξίωμα αυτό πρέπει να έχει γενική εφαρμογή αρχίζοντας από την προταθήσα πρασινοποίηση του πρώτου πυλώνα και το σχέδιο των μικρών γεωργών και καταλήγοντας στις, μετα... στις ρυθμίσεις που έχουν ως αντικείμενο την κοινή στρατηγική με τα άλλα ταμεία, τη σύνδεση με τους μακροοικονομικούς στόχους την ικανοποίηση άλλων εκ των προτέρων όρων και τη δημιουργία αποθεματικού επίδοσης στο δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οι νέες ρυθμίσεις δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγούν σε ομοιρία και καθυστέρηση ως προς την εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ούτε και να διοχετεύουν τους πόρους μονόπλευρα προς τους τομείς που έχουν επιτύχει τους στόχους τους, σε βάρος άλλων εξίσου σημαντικών τομέων. Θέλω επίσης να τονίσω τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε ως Κύπρος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της απάμβλησης της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων και τη δέσμευση άνθρακα. Διαβλέπω όμως μια υποτίμηση ή και υποβάθμιση της τεράστιας προσπάθειας που απαιτείται για την προσαρμογή της γεωργίας και την προστασία των φυσικών πόρων από τις συνέπειες των επερχόμενων αλλαγών. Καταρχήν, η Επιτροπή έχει αποκλείσει την εισαγωγή στα αντικειμενικά κριτήρια κατανομής των πόρων κάποιου κριτηρίου που να σχετίζεται με το μέγεθος της πρόκλησης που συνεπάγεται η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Εκ δευτέρου, δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιηθεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα προέρχεται από την εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές οριακής απόδοσης, όπως αποδεικνύεται εξάλλου με την εμπειρία χωρών όπως η Κύπρος, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις εγκαταλελειμμένης μέχρι πρότινος καλλιεργούμενος γεωργικής γης που υφίσταται κατά έντονο τρόπο τις συνέπειες της διάβρωσης και της απειρήμωσης. Κι όμως οι προτάσεις της Επιτροπής διαφαίνεται να αποκλείουν τις εκτάσεις αυτές αφού δεν τις περιλαμβάνουν στην ενδυνάμει επιλέξιμη γεωργική έκταση με βάση την οποία κατανέμονται εθνικοί φακέλοι. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το πρόβλημα δυνατό να είναι κατά κύριο λόγο μεσογειακό ή περιφερειακό, αυτό όμως δεν δικαιολογεί την παραγνώρισή του. Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω την ανάγκη να υπάρξει το συντομότερο δυνατό περισσότερη διαφάνεια ως προς την κατανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα. Η Επιτροπή έχει αναλύσει στα πλαίσια της μελέσης της αντιχτύπου στις επιπτώσεις διαφόρων υπαλλακτικών σεναρίων και φαίνεται να προσανατολίζεται προς ένα ρεαλιστικό σενάριο κατά το πρότυπο του πρώτου πυλώνα. Εκτιμούμε την προσπάθεια αυτή Θεωρούμε όμως ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ανακοινώσει το ταχύτερο δυνατόν τις προθέσεις της, ώστε να μπορούμε όλοι να τοποθετηθούμε έχοντας υπόψη τη συνολική εικόνα που αφορά την χρηματοοικονομική πλευρά της κοινή γεωργικής πολιτικής. Προσβλέπουμε σε συνέχιση της επικοδομητικής συζήτησης των θεμάτων αυτών και όλων των άλλων και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, κύριο Αλετράρη και θα δώσω τώρα το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Ξεκινάμε με τον κύριο Λουίς ε, Μανουέλ Κάπουλας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, πρόεδρε του Κοινοβουλίου, αξιότιμοι προσκαλεσμένοι, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάλφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσία σας και για αυτή την πρωτοβουλία συμβολίζει την επιθυμία των τριών θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν καλή την πίστη ως συντονιστής ε, του ομάδας των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών και ως εισηγητής. Θέλω να σας εκφράσω, να σας πω ότι η ομάδα μας και εγώ ίδιος είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλες τι υπόλοιπες ομάδες, με το Συμβούλιο και με τον Επίτροπο. Η ΚΑΠ είναι η πιο ε, μια από τις πιο παλιές κοινέ ε, πολιτικέ κοινές και από τις πιο κοινέ, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ε, οι αρχέ τη είναι η εξασφάλιση της ευημερία στην Ευρώπη και η ανάπτυξη του αγροτικού μας δυναμικού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια της κοινής αγροτικής πολιτικής, ιδιαίτερα ε, εν ώψη υπό το φως των εθνικών εγωισμών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στιγμές αυτές είναι δύσκολες. Θα πρέπει ε, όμως, όμως πάντοτε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές προχωράμε και ε, σημειώνουμε πρόοδο. Το έχει αποδείξει αυτό η ιστορία. Θα πρέπει ε, οι ενισχύσεις με δίκαιο τρόπο να κατανεμηθούν ανάμεσα γεωργούς και περιοχές ε, και ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και των φορολογουμένων. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Η ευθύνη μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ε, λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επιδείξουμε ε, πνεύμα διαλόγου. Η Κομισιόν υπέβαλε προτάσεις που ε, σε ό,τι αφορά τις αρχές και τους στόχους τους ε, μας βρίσκουν σύμφωνους εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Κοινοβούλιο ε, έχει ήδη δύο φορές ε, λάβει θέση με σημαντικές ε, πλειοψηφίες εισηγίες των κυρίων Λάιον και Ντες. Τώρα, θα πρέπει οι στόχοι αυτοί και οι αρχές να γίνουν πιο συγκεκριμένα και με αυτόν τον τρόπο να καθησυχάσουμε και τις κριτικές και τις ανησυχίες σε πολλές από τις οποίες είναι και δικαιολογημένες και που έχουν εκφραστεί. Πλευράς προπολογισμού είναι ανεπαρκής ε, σύμφωνα με τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Πολύ δε περισσότερο που το βασικό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, οι άμεσες ενισχύσεις, βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία. Αυτό ε, είναι λανθασμένο. Ε, έχω την εντύπωση ότι η λογική της Κομισιόν είναι τελείως λανθασμένη. Δηλαδή, πρώτα καθορίζονται τα κριτήρια του, των υπολογισμών και μετά οι εθνικοί προϋπολογισμοί σύμφωνα κατά αναλογία μάλλον και βέβαια με την επιφύλαξη ε, διορθωτικών μηχανισμών. Πάντα έτσι συνέβαινε. Γιατί να μην συμβαίνει έτσι, ε, να μην συμβεί έτσι και τώρα. Πάντοτε έτσι ε, συνέβαινε σε όλες τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠΑ. Η άμεση ενισχύση λοιπόν θα είναι το κεντρικό κομμάτι και γύρω από αυτές θα βρεθεί ο συμβιβασμός. Αν λυθεί αυτό το ζήτημα θα βρούμε Συμβιβασμού και στα υπόλοιπα άλλα θέματα. Για το, την, το της ε, ΚΑΠ, ε, το θέμα των μικρών ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των εργαλείων παρέμβασης στις αγορές, τις προτεραιότητες ανάπτυξης πέθρου και στη σχέση ανάμεσα στους δύο πυλώνες και τα διορθωτικά ταμεία. Το η πολιτική μου ομάδα και εγώ ίδιος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας αυτή την ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω και ζητώ και από, τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε, από την Κομισιόν και το Συμβούλιο, ε, να κάνουν το ίδιο. Έτσι ώστε στους ε, επόμενους ε, μήνες να πάρουμε σαφή αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν στο θέμα της κοινή οργανώσεως των αγορών να ξεκινήσω με δύο υπενθυμίσεις. Καταρχήν, ε, όταν, ε, στην έκθεση Albert Des ε, ζητήσαμε την ενίσχυση των παραγωγών στη διατροφική αλυσίδα και προηγουμένως όσον αφορά τη λειτουργία αυτής της διατροφικής αλυσίδας στην έκθεση Μποβέ είχαμε τονίσει ότι μειωνόταν η συμμετοχή των παραγωγών κατά 10% τα τελευταία χρόνια και οι κανόνες της αγοράς δεν μπορούσαν να μας ε, ε, προστατεύσουν από σοβαρές κρίσεις και κανείς δεν μπορούσε να αντιστηθεί. Όσον αφορά τις κρίσεις της αγοράς δημιουργούνται και κλιματικές κρίσεις, υγειονομικές κρίσεις ο, τις οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί γιατί τα περιθώρια κέρδους τους έχουν περιοριστεί με το χρόνο. Άρα υπάρχουν ουσιαστικά θέματα ενδιαφέροντα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να εξετάσουμε, αλλά ε, δεν ε, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό. Δεν πρημοδοτούμε τους παραγωγούς οι οποίοι προσαρμόζονται στην αγορά. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια Πρέπει από κοινού να αναλύσουμε την κατάσταση, να βελτιώσουμε την πρόταση και μου φαίνεται πολύ βασικό να μπορέσουμε να καθορίσουμε από κοινού τους κανόνες ε, της γεωργίας και ε, του ε, θέματος των τροφίμων. Μπορούμε να αφήσουμε να δημιουργούνται τεράστια μαστόδοντα όπως γίνονται στον ανταγωνισμό μας για να δημιουργούνται καρτέλ τα οποία επηρεάζουν και πιέζουν την αγορά. Δεύτερον, η επέμβαση στη λειτουργία της αγοράς ζητά γρήγορη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η αποστολή της και δεν την ε, ξεχνάμε. Πρέπει όμως να σκεφτούμε τις πράξεις κατεξιοδότηση και τις ε, εκτελεστικές πράξεις τις οποίες θέλει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες κατά τη γνώμη μας ανήκουν ε, την ε, διάκριση και λήψη αποφάσεων του Συμβολίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής και κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα το ότι μπορώ σήμερα να συμμετέχω σε αυτή τη συνάντηση γιατί πιστεύω ότι και για μας τους συγητές ε, η μεταρρύθμιση για την γεωργική πολιτική συζητιέται σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή, μια στιγμή όπου μπορεί κανείς να ακούσει όλους ε, τους ε, υπεύθυνο για την κοινή γεωργική πολιτική. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ακούσουμε την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η, η πολιτική γεωργία είναι ιστορική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη πολιτική η οποία συγκέντρωσε τα περισσότερα κονδύλια. Είναι εκείνη η οποία συγκέντρωσε το ίδιο τραπέζι όλα τα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλέξουν σε μια κοινή θέση. Σήμερα λοιπόν είναι σαφής η προστιθέμενη αξία της κοινή γεωργική πολιτικής. Νομίζω ότι όλοι από κοινού μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα επιτύχαναν τα μεμονωμένα κρατημέλη με δική τους εθνική πολιτική. Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης είναι σαφές ότι η γεωργική πολιτική χρειάζεται κονδύλια. Σήμερα λοιπόν στην πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των κονδυλίων που θα διοχετευτούν στη νέα γεωργική πολιτική, εμείς επιμείναμε να υπάρχει ε, μέχρι το 2011 πάγωμα αλλά όσον αφορά τα ε, κονδύλια διαπιστώνουμε ότι θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη μείωση κατά τα επόμενα έτη. Έτσι λοιπόν η μείωση χρηματοδότησης της γεωργικής πολιτικής μέσα στον ευρύτερο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι σαφές ότι η γεωργική πολιτική πρέπει να βαδίζει παράλληλα με το νέο πολιτές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Και αυτό κύριε Επίτροπε, με απασχολεί, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η έγκριση αυτού του νέου πλαισίου μπορεί να γίνει ε, μόνο με ε, ομοφωνία των κρατών μελών. Και επειδή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια βαθιά κρίση, καταλαβαίνετε ότι είναι και διαφορετική η θέση των ε, κρατών μελών. Άρα δηλαδή αυτό είναι κάτι που αναγκαστικά μας ανησυχεί. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθούμε Τη αναθεώρηση, να ασχοληθούμε με το πώ μπορούμε να θεωρήσουμε το κείμενο τη κοινή γεωργικής πολιτική. Να δούμε πώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή. Γιατί αν δεν είναι σαφές ε, το ποια θα είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν για την κοινή γεωργική πολιτική, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του ε, πολιτού χρηματοδοτικού πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος για τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Αυτά δύο πρέπει να είναι σαφές και να συμβαδίζουν. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του ε, χρονοδιαγράμματος, ε, για το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια επιμήκυνση. Είναι απαραίτητο γιατί είναι δύσκολο να ορίσει κανείς τα κονδύλια που θα πάνε για το πρασίνισμα στο πρώτο πυλώνα αν δεν γνωρίζουμε το σύνολο των κονδυλίων. Ή επίσης είναι δύσκολο να ορίσει κανείς την ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική χωρίς να γνωρίζουμε το τελικό ποσό. Είναι δύσκολο να ορίσουμε τους αν δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτή είναι μια διαδρομή, είναι μια πολιτική αν θέλετε που πρέπει να τη χαράξουμε παράλληλα με την αναθεώρηση του πολιτού χρηματοδοτικού πλαισίου. Και υπάρχει ένα πράγμα που με απασχολεί και το προτάσω. Το γεγονός δηλαδή ότι όσον αφορά την προσαρμογή των παλαιών κανονισμών στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, προχωράμε με μεγάλη βραδύτητα στην σύναψη των συμφωνιών. Και έτσι λοιπόν υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης προβλημάτων και θεμάτων. Αυτό όμως δεν είναι θετικό και σίγουρα δεν επιτυχεί τη διαδικασία για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το θέμα της προσαρμογής των κανόνων στη συνθήκη της Λισαβόνας για να καταλήξουμε κατά πόσο ενδεχομένω χρειάζεται κάποια αλλαγή στο περιεχόμενο των κανόνων αυτών. Και κλείνω με μία ευχή ότι το περιεχόμενο χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση τη κοινή γεωρικής πολιτικής μπορεί πράγματι να μας οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των κονδυλίων και μάλιστα και σε αναθεώρηση των κυρωτικών μηχανισμών, οι οποίοι μηχανισμοί αυτοί οδήγησαν στο να εξαιρούνται ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό νομίζω σε σχέση με το παρελθόν πρέπει να αναθεωρηθεί. Βλέπουμε ότι πρέπει κανείς πριν καταλήξει σε συγκεκριμένες περικοπές πρέπει να έχει ε, προβεί σε ανάλυση, σε βαθύτερη ανάλυση των θεμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα προχωράμε με τη συζήτηση. Δύο υπουργοί θα λαμβάνουν το λόγο και μετά δύο ε, βουλευτές. Πρώτον, η Υπουργό, Υπουργός Γεωργίας ε, από το Βέλγιο, η Σαμπρίνα και μετά Υπουργό Γεωργία από το Βέλγιο. Ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής της ε, συνάντησης. Για πρώτη φορά λαμβάνει η χώρα σε αυτό το φορμάτ και είναι μια διαδικασία στην οποία θα πάμε χέρι-χέρι. Είναι η διαδικασία τη συναπόφαση. Δεν θα πω σε λεπτομέρειε, αλλά να πω τα εξή. Να υπογραμμίσω ορισμένα θετικά τη μεταρρύθμιση ε, των προτάσεων. Ε, οι προτάσει ευτυχώ υπάρχουν και μα δίνουν τη δυνατότητα να αρχίσουμε να εργαζόμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεύτερον, ορισμένα μέτρα είναι θετικά. Ιδιαίτερα αυτά για του νέου γεωργού. Ακόμα και αν δεν είναι επαρκή. Επίση, προτάσεις ε, για επίγοντα μέτρα σε περιπτώσεις κρίσεων. Το είδαμε αυτό και στο παρελθόν πόσο σημαντικό είναι. Ε, τρίτον, επιτρέπουν σε οργανώσεις ε, παραγωγών να οργανωθούν και να έχουν έτσι μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Πέρα από αυτά τα θετικά, δυστυχώς υπάρχουν και κάποια αρνητικά από αυτές τις προτάσεις. Κυρίως σε ό,τι αφορά εμάς τουλάχιστον στη δική μας ερμηνεία των κειμένων, στη δική μας ερμηνεία των κειμένων, δεν βλέπουμε πουθενά ούτε απλοποίηση, ούτε αυξημένη διαφάνεια. Αντιθέτως μάλιστα. Ε, έχουμε, είναι σαν λαζάνια αυτές οι προτάσεις, διαφορε, πολλά στρώματα διαφορετικών πραγμάτων σε διαφορετικό πάχος το καθένα μετά η αναδιανομή μεταξύ κρατών μελών και στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους δεν είναι αποδεκτή από εμάς. Για παράδειγμα το Βέλγιο, δεδομένου ότι είμαι υπουργό του Βελγίου, το Βέλγιο θα χάσει ε, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα, παρόλο ότι η γεωργία μας είναι η πιο παραγωγική σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον έχουμε και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που δεν λαμβάνονται υπόψη. Τρίτον, το πρασίνισμα. Ασφαλώς και δεχόμαστε το στόχο, αλλά δεν δεχόμαστε επουδενή τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Είναι υπερβολικά περίπλοκα και δαπανηρά. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Τέταρτον, αρνητικό. Πολύ συγκεκριμένα, η πρόταση για την κατάρριξη του συστήματος ποσοστώσεων στη ζάχαρη από το 2015. Όμω, το, το τη της ζάχαρης ε, μεταρρυθμίστηκε το 2005, βρίσκεται ακόμα σε περίοδο μετάβαση προσαρμογή. Δεν λέμε όχι στην κατάρριξη των ποσοστών ζάχαρης γενικά, αλλά όχι τόσο νωρί. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, και εκεί ε, έχουμε ε, κοινού στόχου, είναι αλήθεια. Ε, έχουμε όμως και διαφωνίες στον ορισμό για παράδειγμα των μηνοκτωσών περιοχών κλπ. Όμως εκεί χρειαζόμαστε πιο τεχνική ανάλυση. Τα κείμενα είναι πολύ τεχνικά, πρέπει να τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο όμως θα χρειαστούμε οπωσδήποτε στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία πολύ πιο συγκεκριμένα ε, που να, στηρίζουν, που να στηρίζουν τις προτάσεις της Κομισιόν με κατανομή ανακράτως μέλος. Και τέλος, μια και πρόκειται για μια πρώτη ανάλυση, ε, λείπει από αυτές τις προτάσεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν βλέπουμε ε, οποιαδήποτε, ε, σα, οποιοδήποτε σαφές μέτρο για την καταπολέμηση της, ε, των ε, μεγάλων διακοιμάσεων των τιμών. Αυτό είναι εις βάρος και των παραγών και των καταναλωτών. Το Βέλγιο βέβαια θα συμμετάσχει όπως πάντα επικοδομητικά και θετικά σε όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Μύροσλαβ Νάγκνχοφ, Υπουργό Γεωργίας από τη Βουλγαρία και μετά θα περάσουμε ε, στους ε, Ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου ε, επιτρέπετε να λάβω το λόγο και να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Γεωργίας και την Προεδρία την Πολωνία όσο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που με ε, κάλεσαν σε αυτή την συζήτηση για τη μελλοντική γεωργική πολιτική. Θα αναφερθώ σε ορισμένες προτάσεις τις οποίες θα σχολιάσω. Καταρχήν, όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, το πρασίνισμα, ε, τις ε, ειδικέ ενισχύσεις και τη συνοχή. Είναι πολύ σημαντικές ε, οι άμεσες πληρωμές για το εισόδημα των γεωργών αλλά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να έχουμε μία χρηματοδότηση ε, επαρκή. Η ανακατανομή μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό μίας, μίας χώρας μέλου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και ελπίζουμε ότι όλοι οι γεωργοί θα μπορέσουν να κριθούν ισότιμα ασχέτως ε, της ε, χώρας τους προελεύσεως. Όσον αφορά αφορά ε, τις, ε, τις ε, άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις ναι μεν είναι ένα βήμα προς τα εμπρός αλλά χρειάζονται και άλλα όσον αφορά τη σύγκληση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα θέλαμε οι πληρωμές να φτάσουν στην κορυφή τους στο 2014 και όχι αργότερα διότι αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση για τους γεωργούς της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας κατά τρόπον ώστε να ε, βρεθούν στη σωστή τους θέση στις ευρωπαϊκές αργορές. Όσον αφορά το πρασίνισμα, η εισαγωγή οικολογικών μέτρων είναι σημαντική ε, αλλά ε, το 30% είναι πολύ υψηλό και χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το ποσοστό για να μπορεί το κάθε κράτος να επιλύει τα οικολογικά του προβλήματα κατά περίπτωση και εξειδικευμένα. Συμφωνούμε ε, με την ε, δυνατότητα να δοθεί βοήθεια σύμφωνα με την ε, πολλαπλή συμμόρφωση, διότι έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε διάφορους τομείς που έχουν προβλήματα, ιδίως για την κτηνοτροφία. Επίσης έχουμε αποθέματα και ε, όσον αφορά το κατόφλι των 150 ευρώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποια ευελιξία και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορέσουν καλύτερα να διαχειριστούν τους σπόρους στα πλαίσια του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα και οι μεταφορές να είναι πιο ευέλικτες. Το έτος αναφοράς το 2011 είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τα προγράμματα που έχουν ε, παρουσιαστεί για το 2014 διότι η Βουλγαρία έχει πιο σημαντικές εκτάσεις από αυτές οι οποίες προβλέπονται, ως εκ τούτου θα χρειαστούμε και περισσότερα προγράμματα. και η τάση αυτή βέβαια θα είναι αυξητική. Όσον αφορά τις επεμβάσεις των αγορών, τις επεμβάσεις στις αγορές, τις διάφορες τομεακές πτυχές, εμείς στηρίζουμε την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων και πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ένα δίκτυο ασφαλείας. Συγχρόνως όμως είμαστε της γνώμης ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα χρειαστεί να ληφθούν όσον αφορά την, την ανάπτυξη της υπαίθρου και τις προτελεότητες, ε, του στόχους και τα πακέτα για την αξιολόγηση του κινδύνου. Εμείς στηρίζουμε όλα τα μέτρα τα οποία τίνουν σε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ του γεωργικού και δασοκομικού τομέα, ε, όπως επίσης ε, του επαγγελματικού επαγγελματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την περικοπή 5% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τήρουμε τον χρόνο που έχει προβλεπτεί ε, έχοντας κατά νου και κάποιους ε, συναδέλφους που ε, είναι αναγκασμένοι να φύγουν πριν τελειώσει η συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Άλμπερτ Ντες. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίε Υπουργοί από τα κράτη-μέλη, ε, κυρίες και κύριοι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβαν μια τεράστια ευθύνη για τη γεωργική πολιτική του 2013. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση για 14 εκατομμύρια γεωργούς οι οποίοι καλλιεργούν πάνω από 170 εκατομμύρια εκτάρια. Έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πρέπει να ε, έχουν κάθε μέρα φρέσκα προϊόντα και έχουμε εν πάση περιπτώσει ευθύνη για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια θέσεων εργασίας στη Γεωργία. Αν δούμε λοιπόν τι συνέβη στην Ευρώπη κατά τις ε, τελευταίες ε, δεκαετίες ε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν εξίσου προβλήματα όπως και σε άλλους τομείς. Αν δούμε λιγάκι τα στοιχεία θα δια... ίσως πει κανεί ότι τα μεγαλύτερα ελλείμματα τα έχει η ορική πολιτική. Δεν είναι αλήθεια όμως, αλλού υπάρχουν τα ελλείμματα. Σε ε, πάρα πολλούς ε, τομείς. Οι πολιτικοί σκέπτονται μόνο από τη μία εκλογική περίοδο στην άλλη. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ε, δεν θέλω, δεν επιθυμώ να προτείνονται μέτρα τα οποία περιορίζουν τα δικαιώματα των γεωργών. Διάβασα κύριε Επίτροπε τις περισσότερες από τις 650 σελίδες την προηγούμενη εβδομάδα το έκανα αυτό και τρόμαξα γιατί αποκόμισα την εντύπωση ότι στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυξάνεται το γραφειοκρατικό άκτος. Ε, κύριε Επίτροπε, συμφωνώ μαζί σας ότι πριν επικρίνουμε θα πρέπει πρώτα να διαβάσουμε όλες τις προτάσεις. Και εγώ πιστεύω ότι όταν κανείς ε, επικρίνει ή καταθέτει κριτική θα πρέπει να καταθέτει παράλληλα και τις αντιπροτάσεις του. Γι' αυτό λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ως Υπουργοί έχουμε χρονικό διάστημα πράξουμε αυτό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι στις προτάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, διαβάν, δεν λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το 2013 πρέπει η Γεωργία να έχει καλές ε, προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ελλείμματα όπου ε, δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θέλω το να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι το γνωρίζουν. Ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και γι' αυτό κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να ασχοληθούμε σε βάθος με τις ε, προτάσεις. Η χρηματοψηφιακή κρίση έχει οδηγήσει και στο ότι η γεωργία δικοί μας ε, έχουν λιγότερα χρήματα και έχουν αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος. Εμείς δεν θα το δεχτούμε αυτό. Εμείς θα αντισταθούμε έτσι ώστε οι γεωργοί μας να έχουμε προοπτικές στο μέλλον. Και εσείς κύριε Επίτροπε αλλά και όλοι οι υπόλοιποι έχουν το καθήκον η πολιτική να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι προτάσεις που κατατίθενται να είναι και εφαρμόσιμες στην πρακτική για τους γεωργούς. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Η σημερινή συνάντηση πιστεύω ότι ε, μπορεί να δώσει την ευκαιρία να ανταλλαγούν απόψεις ε, ανάμεσα στους Υπουργούς Γεωργίας των κρατών μελών αφενός υπουργοί οι οποίοι έχουν άποψη, έχουν αξιολογήσει τις προτάσεις Κομισιών και τους ευρωβουλευτές αφετέρου. Οι ευρωβουλευτές και οι οι υπουργοί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή, έχουν ξανασυζητήσει ε, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, αλλά είναι πολύ σημαντικός και ο σημερινός διάλογος. Οι απόψεις του Κοινοβουλίου που έχουν εκφραστεί σε παλαιότερες γνωμοδοτήσεις εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά το μέλλον της ΚΑΠ. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ε, απορίες ε, σε, για διευκρίνηση στα σημεία των προτάσεων. Σε, ό,τι αφορά, σε όμως τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο έχει πει ότι δεν θα δεχτεί καμία περικοπή του προϋπολογισμού της γεωρικής πολιτικής. Διότι αν συμφωνούμε για τις προκλήσεις, αν συμφωνούμε για τα προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν, αν συμφωνούμε για το ποια πρέπει να είναι τα εργαλεία και οι πολιτικές που χρειαζόμαστε, πρέπει να συμφωνήσουμε και για έναν επαρκή προπολογισμό. Μετά υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία ορισμένοι ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει ε, αμφιβολίες και διαφωνίες επιφυλάξεις. Ε, ο Επίτροπος είπε ότι η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη την ε, ποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια αυτό, σε ορισμένε τυχές τουλάχιστον. Για παράδειγμα, έχουμε ε, ε, ενιαίες ενισχύσεις ε, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία των περιπτώσεων και καταστάσεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πιστεύω ε, ότι θα πρέπει οι προτάσεις αυτές να προσαρμοστούν περισσότερο. Ε, υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που θα ήθελα να θίξω, αλλά θα θίξω μόνο ένα ακόμα, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο Επίτροπος είπε σήμερα ότι θέλει να διατηρήσει την παραγωγή σε όλες τις περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η περίπτωση της ζάχαρης είναι μια πολύ σαφής περίπτωση που μια κακή ε, ε, απόφαση οδηγεί σε εγκατάλειψη της παραγωγής σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλύτερα, να μελετήσουμε πολύ περισσότερο τις προτάσεις της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τι ποσοστώσεις της ζάχαρης που επιθυμεί να καταληφθούν μέχρι το 2015. Το Κοινοβούλιο έχει ε, ήδη πάρει θέση, αντιτίθεται σε αυτό. Είναι ζητήματα στα οποία θα πρέπει να βρούμε μια σύγκληση, να ανταλλάξουμε απόψεις και να κάνουμε μια πρόταση που θα εγγυάται τελικά το μέλλον του τομέα, ε, τη βιωσιμότητά του και την παραμονή των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές, κάτι που αυτή τη στιγμή ε, διακινδυνεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που λαμβάνει η χώρα αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι θα βοηθήσει τον γεωργικό μας κόσμο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα θα να δώσω το λόγο σε δύο υπουργού, ε, στην Υπουργό ε, της Γερμανίας και στην Υπουργό της Ισπανίας κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά που με καλέσατε να συμμετάσχω στη σημερινή συνεδρίαση, ε, την κοινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής ε, του Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ε, Συμβουλίου των Υπουργών. Θα ήθελα επίσης εξ αρχής να σας πω ότι η Γερμανία στηρίζει τους σημαντικούς στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως το είπαν ορισμένοι συνάδελφοι και εμείς θεωρούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Εν ευθέτω χρόνο. Και εγώ θα ήθελα σήμερα να αφαιρθώ σε ορισμένα εξ αυτών. Καταρχήν βλέπουμε ότι η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακατανομή ε, του όγκου των άμεσων ενισχύσεων είναι ένα διαφανές σύστημα και το χαιρετίζουμε αυτό. Όμως ε, χρειαζόμαστε διαφάνεια όσον αφορά το σύνολο του προβλησμού, δηλαδή ε, τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, χρειαζόμαστε την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων ανάμεσα στα κρατημέλη. Αυτό θα αποφασιστεί από κοινού με το μέλλον των ενισχύσεων και σε σχέση και με άλλους τομείς της ε, γεωργίας όπως είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου και τα διαρθρωτικά ταμεία. Πράγματι, ε, χρειαζόμαστε μία ανακατανομή των ε, άμεσων ενισχύσεων. Εμείς στη Γερμανία έχουμε κάνει πολύ καλή εμπειρία σχετικά με το θέμα αυτό. Όσον αφορά η ο συσχετισμός των άμεσων πληρωμών με την ε, υποκαλλιέργεια ή την καλλιεργούμενη έκτεση, αυτό δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Στην ε, Γερμανία λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της μισθοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιθυμεί μάλλον να αποκόψει πλήρως την παραγωγή από τις άμεσες ενισχύσεις. Εμείς επιθυμούμε να ξεκολουθήσει να ισχύει αυτός ο συσχετισμός, έστω και αν θέλετε για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα. Δεύτερον, όσον αφορά τις ε, συνεισφορές για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Γερμανία θεωρεί ότι πράγματι πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω οι συνεισφορές αυτές. Τούτο όμως πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τους στόχους ε, της ε, παροχής ε, τροφίμων και σε σχέση με την χρήση πρώτων υλών. Βεβαίως πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι ήδη σήμερα η γεωργία συμβάλλει σημαντικά για την επίτευξη των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος. Οι γεωργοί οι οποίοι ήδη σήμερα συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση αν υπάρξει περαιτέρω πρασίνισμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η εξαίρεση των οικολογικών ε, καλλιεργιών από το πρασίνισμα στον δεύτερο πυλώνα. Τρίτον, ανάπτυξη της υπέτρου για τα μέτρα ενίσχυσης και για την ενίσχυση της υπέτρου χρειαζόμαστε την ασφάλεια. Δεν πρέπει να υπάρξει άμεση αλλαγή και απότομη αλλαγή των κονδυλίων που χορηγούνται στα κράτη-μέλη. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ένας ε, διαχωρισμός ε, με τις ε, μειονεκτούσες περιοχές. Εμείς επιθυμούμε να διατηρήσουμε τον σύστημα των μειονεκτουσών περιοχών που έχουμε στη Γερμανία. Όσον αφορά τώρα τις ε, συμφάσεις, ε, συμβάσεις ε, συνεργασίας, κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τελευταίο σημείο που είναι πολύ σημαντικό για μένα, στην απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η απλούστευση αυτή είναι καθοριστική σημασία για μας και γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προχωρήσει περαιτέρω με τη μεταρρύθμιση γιατί η προσέγγιση που έχει τώρα δεν αρκεί. Σε γενικές γραμμές θέλω να πω ότι ε, κατά την άποψή μας δυστυχώς αυτές οι προτάσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των δαπανών. Τελειώνοντας όμως θέλω να πω ότι και εγώ θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά διαδικασία και το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν και πρέπει να βρουν καλές λύσεις για να υπηρετήσουν την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Ρόζο Αγγιλάρ ξέρετε, αλλάζω λιγάκι τη σειρά των Υπουργών, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πρέπει να ε, τηρήσω και ε, την αναχώρηση των ε, πτήσεων. Η κυρία Ρώσα Αγγιλάρ, Ριβέρο από την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω αυτούς που διοργάνωσαν την συνεδρίαση αυτή Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική, πολύ θετική, αποτελεί ένα βήμα διαλόγου, ε, απολύτως απαραίτητο. Η Ισπανία θέλει να είναι επικοδομητική και ταυτόχρονα ε, θα εκφράσουμε με απόλυτη σαφήνεια τη θέση μας. Η Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η γεωργία είναι στρατηγικός κλάδος με σαφή ε, στόχο την τροφιμική επάρκεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία έχει θέση, κοινή θέση με όλες τις αυτόνομες περιοχές της, ε, θέση την οποία στηρίζει όλος ο τομέας, όλος ο κλάδος μέσω των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους αγρότες και τους παραγωγούς. Με αυτή την έννοια η θέση μας είναι η Οι προτάσεις Κομισιόν δεν έλαβαν υπόψη επαρκώς τις απόψεις μας που εξέφρασε η υπουργό μας ε, για, το θέμα, για, τα θέμα, για το θέμα της μεταρρύθμισης ΚΑΠ επανειλημμένος. Ε, εμείς διαφωνούμε κυρίως με το θέμα της, των άμεσων ενισχύσεων, διότι οι προτάσεις Κομισιόν δεν αναγνωρίζουν τις διαφορετικές καταστάσεις, τις διαφορετικές ζώνες και μεθόδους παραγωγής με αυτόν τον τρόπο, με τις προτάσεις της Κομισιόν, θέτει σε κίνδυνο ε, ένα μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα τις πιο ε, παραγωγικές, ε, τις πιο αποδοτικές, που έχουν όμως και το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Η πληρωμή μιας ενίας ενίσχυσης θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε μεγάλο το κομμάτι του τομέα. Ε, πολύ δε περισσότερο που με αυτόν τον τρόπο χάνει την κοινωνική της, ε, ε, τον κοινωνικό της λόγο ύπαρξης. Ε, σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα της ΚΑΠ, συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι κάνουν ήδη οι γεωργοί μας, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις, με τις περιβαλλοντικές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη. Δηλαδή, δεν ξεκινάμε από το μηδέν, η γεωργή μας ήδη εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα, διατάξεις και κανόνες στους οποίους θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δεν πρέπει να θίξουμε την την παραγωγικότητά τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Δεν συμφωνούμε επίσης με τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Θα πρέπει ο ορισμός αυτός να βελτιωθεί πολύ. Η πρόταση επίσης απλούστευσης της ε, ΚΑΠ ε, καταλήγει να <laughs> είναι το ακριβώς αντίθετο η ΚΑΠ γίνεται πιο περίπλοκη και πιο γραφειοκρατική για τον Γεωργό και τον παραγωγό. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τη διαχείριση αγοράς, ε, χρειαζόμαστε εργαλεία που να είναι χρήσιμα, αποτελεσματικά και ευπροσάρμοστα, ε, να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα και γρήγορα στις αλλαγές στις αγορές, στις διακυμάνσεις των τιμών και σε περίοδους κρίσης. Επίσης, θα θέλαμε να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητα με τρόπο πολύ καθαρός προτάσεις έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ανταγωνιστικότητας για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με τρίτες χώρες με τις οποίες μπορούν να συναυτούν συμφωνίες. Επίσης, μια άλλη αρχή που είναι πολύ σημαντική είναι η αρχή της ισορροπίας της τροφιμικής αλυσίδας. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών έτσι και ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι κανόνες ανταγωνισμού. Συνεπώς, οι προτάσεις που έχουν γίνει θα πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες προτάσεις. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα της ανάπτυξης πέθρου, επουδενή δεν θα πρέπει ο, το ποσοστό συγχρηματοδότηση να είναι πάνω από 50%. Η πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου θα πρέπει να λάβει υπόψη την κατάρτιση την και την καινοτομία ως βασικά στοιχεία της και θα πρέπει ταυτόχρονα να διατηρήσει τις επενδύσεις σε υποδομές, ε, σε άρδευση έτσι ώστε ο αγροτικός πληθυσμός να παραμείνει στην Ήπεθρο, να βελτιωθεί η ζωή του και οι προσδοκίες του να ικανοποιηθούν. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν να αυξήσουμε τον αριθμό των γεωργών. Το 2% του, πρώτου, του προπορισμού του πρώτου πυλώνα ε, που έχει προβληθεί για τέτοιου είδου ε, μέτρα είναι ανεπαρκές. Θα πρέπει να πείσουμε τους νέους ε, Ευρωπαίους ότι έχουν μέλλον στη γεωργία και ότι έχουν χώρο στη γεωργία για να αναπτύξουν εκεί την επαγγελματική και την προσωπική του ζωή. Συνεπώ, ο δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετα μέτρα για του νέου γεωργού και μέτρα στήριξης των γυναικών στην γεωργία και στην ε, Ήπεθρο. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια πρόταση για ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που δεν κάνει ούτε μία αναφορά στη γυναίκα, με δεδομένο το ρόλο της γυναίκας σε αυτές τις περιοχές και στη γεωργία. Γι' αυτό το λόγο αρχικά είχαμε απορρίψει τις προτάσεις της Κομισιόν. Διότι πέραν των όσων είπα, βλάπτει το παραγωγικό μοντέλο όχι μόνο της Ισπανίας, αλλά και Τη γεωργίας όλων των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση, οι οποίες δεν λαμβάνονται παρκώ υπόψη. Δεν λαμβάνονται παρκώ υπόψη η Μεσόγειος ε, με όλη την ποικιλία και τον πλούτο της. Ε, τώρα το λόγο ε, θα λάβουν οι βουλευτές. Πρώτα θα λάβει το λόγο ο George, George Lyon. Ευχαριστώ πρόεδρε και επίσης ευχαριστώ των Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να μπορούν να συναντηθούν και να συνεδριάσουν οι τρεις ε, θεσμοί. Η παραγωγή των ε, τροφίμων και η τροφιμική ασφάλεια ποτέ δεν ήταν πιο σημαντική από ό,τι βλέπουμε τώρα. Τώρα υπάρχει μεγάλη διακύμανση των τιμών και το έχουμε συζητήσει αυτό επανειλημμένα. Έχουμε πει ότι ε, δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός, ε, μειώνεται η παραγωγή τροφίμων, υπάρχει λειψιδρία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις επηρεάζουν τους ε, γεωργούς. Και όσον αφορά το βασικό ερώτημα, το κατά πόσον οι μεταρρυθμίσεις ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ε, προκλήσεις, κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ένα νέο μοντέλο περισσότερο αποτελεσματικό από πλευράς ενέργειας και εκπομπών διεξιδίων του άνθρακα, η απάντηση είναι δυστυχώς όχι, ως έχουν τα πράγματα. Υπάρχει βέβαια μία πολύ καλή αρχή, όμως δεν δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες για μια περισσότερο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία. Θεωρώ ότι καλά στοιχεία είναι το ότι προβλέπεται δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων, παρότι θεωρώ ότι ορισμένα κρατημέλη πιστεύουν ότι αυτή η πρόταση δεν προχωράει αρκετά. Να υπάρχει καλύτερη κατανομή ε, και ανάμεσα στους ε, γεωργούς ε, πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να αφήσουμε το παραδοσιακό μοντέλο ε, και να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο ε, πληρωμών. Επίσης, εκείνο που χαιρετίζω είναι οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Πολύ σημαντικές αυτές οι επενδύσεις ε, στο μέλλον. Θα είναι στο μέλλον. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα ορίσουμε και τις άμεσες πληρωμές οι άμεσες πληρωμές. Τι θα γίνει με τις πληρωμές αυτές ε, στις ε, μειονεκτούσες περιοχές. Εκείνο που χαιρετίζω επίσης είναι η έννοια του πρασινίσματος των άμεσων ενισχύσεων. Το Κοινοβούλιο το ζήτησε αυτό σε δύο περιπτώσεις και εμείς επιθυμούμε να στηρίξουμε αυτή την έννοια. Αλλά αυτό που υπάρχει εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι οι λεπτομέρειες. Γιατί νομίζω ότι ε, τα μέτρα έχουν σχέση με την ε, περίφημη cross-compliance ε, και αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχουμε μέτρα περισσότερο αποτελεσματικά ουδέτερα ως προς την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Οι ε, προτάσεις λοιπόν αποτελούν μια πολύ καλή αρχή. Ελπίζω οι θεσμοί να συνεργαστούν για να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα, να έχουμε ένα νέο μοντέλο που είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον ε, και θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, γίνει μια βελτίωση στο μέλλον αν όλοι προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τότε είμαι σίγουρος ε, ότι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και θα μπορέσουμε να ε, διασφαλίσουμε την διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού. Αντιπρόεδρος Βατσεβόσκη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν πολλά θετικά στιμία στις προτάσεις που είναι στο τραπέζι σχετικά με τους ενεργούς ε, γεωργούς, το πρασίνισμα, τη στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων, αλλά είμαι ο μόνος σκιώδης εισηγητής για τις άμεσες ενισχύσεις και άμεσες πληρωμές που προέρχεται από τα νέα κράτη και γι' αυτό θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με τον ισοσκελισμό των αμέσων πληρωμών. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων κρατών παρόλο που αυτό δεν ισχύει πάντοτε διότι υπάρχουν και μικρές άμεσες πληρωμές σε παλιά κράτη-μέλη αλλά όταν ε, ανέφερα στην Πολωνία κοινωνία το σύστημα αυτό του, είπα ότι έχω και καλά νέα και κακά νέα δηλαδή ότι θα καταργηθούν οι άμεσες πληρωμές αλλά δεν ξέρουμε πότε. Και εδώ, εφόσον δεν υπάρχουν εκπρόσωποι της Δανίας εδώ, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα παλαιού και νέου κράτους. Δεν θα αναφερθώ στην Πολωνία, γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσω ένα διαφορετικό παράδειγμα, τη Λιθουανία και τη Δανία, ένα παλιό και ένα νέο κράτος μέλος που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος σε ε, δύο ε, είναι και οι δύο χώρες της Βαλτικής και έχουν ε, παρεμφερεί σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στο παράρτημα 2 μιλάμε για τις άμεσες πληρωμές οι οποίες θα αποδοθούν στα κράτη αυτά. Το 2013 η Δανία θα λάβει 942 ε, ε, εκατομμύρια και ε, η Λιθουανία 342. Δηλαδή όταν θα σταματήσει αυτή η εξισορρόπηση. Η διαφορά θα είναι Δανία 909 και ε, η Λιθουανία 458, δηλαδή το ίμιση. Γιατί λοιπόν υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Η Δανία είναι μήπως μία ορεινή χώρα, όχι βέβαια, οι καταστάσεις ε, είναι ακόμη πιο ίσες ε, και τέλειες από ό,τι στην Λιθουανία. Η Δανία δεν χρειάζεται να καλύψει το χαμένο χρόνο από την ε, κομμουνιστική εποχή. Η Λιθουανία το χρειάζεται. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο διπλασιασμός των ε, αμέσων πληρωμών. Απλώς η απάντηση είναι διάκριση. Διάκριση η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 18 της ε, συνθήκης που κατήρτισε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μου αρέσει να μιλάμε για βαθμιαία ισοπαίδωση των διαφορών, διότι αυτό είναι κάτι που ισχύει από το 2004. Ξεκινήσαμε με δεσμενέστερες συνθήκες και κάποια στιγμή έπρεπε να φτάσουμε το, στο ίδιο επίπεδο αμέσων πληρωμών που έπρεπε να έχουν εξισωθεί το 2013. Πόσο χρόνος θα χρειαστεί. Δεν συνάδει αυτό με τις αρχές Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν λύνει το πρόβλημα διότι η ε, καταβολή αμέσων πληρωμών είναι πολύ σημαντική για την γεωργία αν θέλουμε να έχουμε παντού γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε μερικά σημεία μόνο. Δίνουμε το λόγο στον Υπουργό της Τσεχίας ε, και κατόπιν ε, στον Υπουργό της Πορτογαλίας. Πρώτα απ' όλα στον Υπουργό της Τσεχίας, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου Λομιλτής, κυρίες και κύριοι, ε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να ε, μπορώ να συζητήσω μαζί σας, να έχω αυτή την παρέμβασή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι αλλάξατε τη σειρά των ομιλητών, αν ήμασταν στην Τσεχία, στην Τσεχία λένε ότι προηγούνται οι κυρίες και προφανώς ισχύει αυτό και εδώ. Από ό,τι είδα προηγήθηκαν οι κυρίες. Δεν πειράζει. Τώρα λοιπόν θα πω μερικά λόγια για αυτά τα οποία μας απασχολούν. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω και εδώ ότι όσον αφορά την Τσεχία είναι σημαντικό η νέα γεωργική πολιτική ε, να είναι διαφανής ε, και να μην συνεπάγεται μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος. Βεβαίως και να είναι και ανταγωνιστική. Δυστυχώς ορισμένες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν μας προβληματίζουν. Ε, θα ήθελα να πω ε, κάτι για ορισμένα θέματα που ετέτσαν. Καταρχήν όσον αφορά τις ε, άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται στους γεωργούς. Στο μέλλον οι άμεσες ενισχύσεις δεν θα αποτελούν απλούστευση. Τουναντίον θα συμβαίνει Ακριβώς το αντίθετο. Ε, γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υπέρ του ισχύοντος συστήματος που προβλέπει την ενισχύση με σημείο αναφορά την καλλιεργούμενη έκταση, τα εκτάρια. Ε, και επιθυμούμε ε, αυτό το σύστημα να διαρκέσει μέχρι το 2020. Και η οικολογικοποίηση, όπως λέγεται, των πληρωμών, καλή και αυτή, αλλά να είναι προαιρετική. Και το ύψος των πληρωμών εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής της κοινή γεωρικής ε, πολιτικής. Ο κύριος ε, Επίτροπος ε, είπε ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ευρώπη. Εκείνο που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι η παραγωγή. Συμφωνούμε μαζί του. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η πρόταση του 7% αυτή η πρόταση είναι αντίθετη με την ε, προαναφερθήσα τάση και γι' αυτό λοιπόν επιθυμούμε η Κομισιόν να καταλήξει σε μια καλύτερη ε, πρόταση. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευελπιστούμε, θέλουμε να υπάρξει συμβιβασμός και αυτό το είπα και στο τελευταίο συμβούλιο. Η πρόταση που έχει κατατεθεί εμάς δεν μας αρέσει. Όσον αφορά τις ε, άμεσες ενισχύσεις, θέλουμε να σας πούμε ότι η Τσεχία τάσεται κατά οποιασδήποτε μορφής μέτρων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα αντικειμενικά κριτήρια και το ανώτατο όριο. Και εδώ θεωρούμε ότι θα προκύψει μεγαλύτερη γραφειοκρατία στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό διαφωνούμε. Όσον αφορά τώρα την πρόταση για την ανάπτυξη του ε, δεύτερου πυλώνα. Εμείς αυτό το θεωρούμε καθοριστική σημασίας θέμα και πιστεύουμε ότι τα κονδύλια για την ανάπτυξη της ε, υπέτρου, τα κονδύλια αυτά οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα κάθε κράτους μέλους και αυτό να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό. Ε, στηρίζω την κυρία Καρσία Περές ε, σε αυτό που είπε ότι το, Ευρωπαϊκό, το Κοινοβούλιο θα είναι αντίθετο με περικοπές σε αυτό το τομέα. Αυτό με καθιστά αισιόδοξο. Το νέο χρηματοδοτικό ε, πλαίσιο θα αφορά και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε και για τα κονδύλια που θα συνοδέψουν αυτό το πλαίσιο. Ε, θα υπάρξει εναρμόνιση των κανονισμών. Οι συμβάσεις ε, που βασίζονται στην αιρεσιμότητα, εμείς αυτές τις απορρίπτουμε και πιστεύουμε ότι ε, η υποστήριξη της υπέτρου πρέπει να γίνει με σημείο αναφοράς την αναγκαιότητα και το κράτος μέλος. Εμείς θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνεται η παραγωγή και η ζωή στην Ήπετρο και δημιουργούνται και θέσεις ε, εργασίας. Ε, τελειώντας, ε, θέλω να πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την άποψη της Τσεχίας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα που την άποψή μου δεν την παρουσίασα μόνο στους βουλευτές αλλά και στον Επίτροπο και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και στο μέλλον. Η Πορτογαλίδα Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα σε αυτή την τριμερή συνάντηση Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εντάχει την θέση της Πορτογαλίας για τα κεντρικά ζητήματα των προτάσεων της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές, η Πορτογαλία συμφωνεί με τον ε, στόχο σύγκλησης με τις ε, εθνικές πληρωμές, μεταξύ των εθνικών πληρωμών. Όμως, ε, αυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα και στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών. Υπ' αυτή την έννοια, οι προτάσει τη Κομισιόν δεν είναι δίκαιε ούτε και επαρκεί. Το κριτήριο, άλλωστε, θα πρέπει να είναι το ίδιο και για μας θα πρέπει να είναι το κριτήριο της χρησιμοποιούμενης γεωρικής έκτασης. Σε ό,τι διαφορά το πρασίνισμα της ΚΑΠ, ε, η Πορτογαλία θεωρεί θετικό το πρασίνισμα για την βιωσιμότητα της γεωργίας. Όμως, θα πρέπει να προσαρμόσουμε καλύτερα την πολιτική μας και να την κάνουμε πιο ευέλικτη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών και ιδιαίτερα τις ιδιαιτερότητες των μεσογειακών καλλιεργιών. Η εισαγωγή ενός εθελοντικού χαρακτήρα του πρασινίσματος είναι θετική. Ε, Ω κριτήριο επιλεξιμότητας επίσης θα μπορούσε να ε, επιλεγεί αυτό που έχει επιλεγεί και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη και στην Πορτογαλία σε ό,τι αφορά την χρήση των περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τους, τους ε, μικρούς γεωργούς και τα μέτρα της απλοποίησης θεωρούμε πολύ θετικές προτάσεις Κομισιόν. Ε, ό,τι αφορά τους ενεργούς ε, γεωργούς και τον ορισμό τους, ε, θεωρούμε ότι το πρώτο σημείο για το 5% είναι υπερβολικά περίπλοκο, πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Αλλά το δεύτερο κριτήριο που έχει σχέση με την ε, μη εγκατάλειψη είναι πολύ καλό και δίνει το μήνυμα ότι οι γεωργοί θα πρέπει να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεσμεύεται υπέρ μιας γεωργίας που ε, θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα των τροφίμων στα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ε, των αγορών, δύο πράγματα. Όπως και άλλα κράτη-μέλη, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πάμε πιο μακριά στην λειτουργία της τροφιμικής αλυσίδας, ε, αναζητώντας ε, καλύτερου μηχανισμούς για την καλύτερη κατανομή της αξίας. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την ε, διατήρηση των ποσοστώσεων γάλατος και το καθεστώς των δικαιωμάτων φύτευσης στην, στον, ε, τομέα του ίνου. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνου, οι προτάσει Κομισιόν είναι καλέ και πολύ σημαντικέ ε, για χώρε όπω η Πορτογαλία, ε, που χαρακτηρίζονται από κλιματική αστάθεια. Τα μέτρα για τι οργανώσει παραγών είναι επίση θετικά, παρόλο ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάμε πιο μακριά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις ε, προσπάθειες ε, οργανώσεων που ήδη υπάρχουν. Τέλος, για πολύ συγκεκριμένα μέτρα που επηρεάζουν την Πορτογαλία, το θέμα των επενδύσεων, για παράδειγμα, στην άρδευση, για χώρες όπως η Πορτογαλία που ε, υφίστανται ε, το αποτέλεσμα ξηρασίας πολύ συχνά, αλλαγή κλιματικών ε, μεταστροφών και αλλαγών, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε επενδύσεις στην άρδευση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί η γεωργία να γίνει και πιο βιώσιμη. Τελειώνω λέγοντας ότι χειροκροτούμε, επικροτούμε μάλλον την Κομισιόν για την σημασία που δίνει στην ΚΑΠ. Μια ισχυρή ΚΑΠ που θα ε, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της επάρκειας των τροφίμων στο μέλλον και που θα καθιστά την ε, Ευρώπη σημαντικό παίκτη παγκοσμίω. Ευχαριστώ πολύ. Vă mulțumesc. Trebuie să menționez că mi-am permis să-i dau cuvântul doamnei ministru în, înaintea ordinei stabilită pe lipsă. Pe... lipsă εις ε, την ε, Υπουργεία ε, ο κύριος Χόισλινγκ. Κυρίες και κύριοι, η αναθεώρηση για την πολιτική μας ομάδα βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση διότι σύμφωνα με τους ε, ευρωπαϊκούς κανόνες ε, συμμορφώνεται, βασίζεται σε μία στρατηγική βιοπικιλότητος και αυτή θα είναι η μελλοντική πολιτική ε, και γι' αυτό θέλουμε η παραγωγή να βασίζεται σε ποιότητα, και εις ε, την περιφερειακή ε, παραγωγή. Λέγεται από τη μία πλευρά ότι ε, πρέπει να παράγουμε περισσότερο, αλλά όταν πετάμε το 50% των τροφίμων που δεν καταλήγουν στο πιάτο μας, πρέπει να αναρωτηθούμε αν όντως πρέπει να επικεντρωθούμε στην αύξηση της παραγωγής, διότι όπως πολύ σωστά λέχθηκε για πολλά μέτρα πιστεύω ότι το να τίνουμε σε μη, στο 70% δεν είναι η σωστή λύση και ενώ έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές για το πρασίνισμα τώρα κολλάμε στις λεπτομέρειες πρέπει να ε, γίνει αποδεκτό και από τους πολίτες και από τους φορολογούμενους και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις δύο πτυχές. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να δούμε πώς ε, θα εμπλακούν οι δημόσιοι πόροι. Ε, επίσης, το θέμα της υπεράσπισης δεν έχει και της κατανομής δεν έχουν επιληθεί με ε, ένα ε, πλαφόν 120 δισεκατομμυρίων δεν ε, επιτυγχάνουμε και αυτή τη στιγμή ε, οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις είναι αυτές οι οποίες πρημοδοτούνται. Πρέπει να βελτιώσουμε και την διατροφική αλυσίδα και εδώ αναφέρομαι στο θέμα του γάλακτος. Πιστεύω ότι το θέμα του γάλακτος πρέπει να ξανασυζητηθεί. Χρειαζόμαστε νέους κανόνες όχι μόνο στους τομείς κρίσεως αλλά παντού διότι έχει αποτύχει η πολιτική μας και είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να ενισχυθούν και οι γεωργοί στην αλυσίδα. Όσον αφορά τους ενεργούς γεωργούς, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες. Χρειαζόμαστε βέβαια μία στρατηγική των λευκομάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εισάγει ένα μεγάλο ποσοστό. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Όσον αφορά την ευελιξία και τους πυλώνες δεν είμαι αντίθετο στην ευελιξία αλλά θα πρέπει να αναφερθεί αυτό και στο δεύτερο πυλώνα και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και να υπάρχει ισορροπία. Πολλά ελέγχθησαν και θέλω να κάνω μία έκκληση στους Υπουργούς Γεωργίας οι οποίοι πρέπει να προβλέψουν επαρκή χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής διότι άλλωστε τα κράτη-μέλη πρέπει να τροφοδοτήσουν τον προϋπολογισμό για να έχουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική που να αξίζει το όνομα ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα και μία πολύ αποδοτική συζήτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Τσόλος, ο οποίος λέει ότι συναντιόμαστε συχνά και συζητάμε, ιδίω όσον αφορά την πολιτική που θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί μέχρι το 2020. Δεν ακούω όμως όλα αυτά για πρώτη φορά και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε δημιουργηθεί μία κατάσταση όπου πολλά λέμε, πολλά υποσχόμεθα, ε, αλλά στο τέλος όταν βλέπουμε τους ουσιαστικούς αριθμούς τότε ε, δεν ε, ικανοποιούμαστε και δεν έχουν καμία σχέση οι αριθμοί με αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή δεν ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές συνθήκες οι οποίες αυτή τη στιγμή προβλέπονται στην κοινή γεωργική πολιτική, ιδίω στις ε, μικρές επιχειρήσεις, τους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση. Στη χώρα μου, στην Λετωνία διότι εγώ είμαι ε, βουλευτής από τη Λετωνία ε, το θέμα που μας απασχολεί είναι οι άμεσες ενισχύσεις διότι αν σήμερα η Λετωνία αλλά και η Λιθουανία και η Εσθονία παίρνουν μόνο το 30% της μέσης τιμής των ενισχύσεων ενισχύσεων μας λέγουν «Ε, γιατί ενοχλείστε μέχρι το 2 2020 θα έχετε 50% αλλά ήδη θα είμαστε πέραν των 15 ετών μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν νομίζω ότι οι λετωνοί πολίτες θα χαρούν πάρα πολύ να στηρίξουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις προσπάθειές του. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε. Όταν κάποιος λέγει ότι δεν υπάρχουν πόροι, εγώ ρωτώ αυτό που μου με ρωτούν και οι ψηφοφόροι μου ε, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμυρίων επενδύσεις για να ε, γίνει ποδηλατοδρόμιο όπως αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο γιατί υπάρχουν πόροι που εξαφανίζονται σε μία μαύρη τρύπα ε, νομίζω κύριε Επίτροπε ότι πρέπει να απαιτήσετε περισσότερα όταν αυτά συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον κύριο Μπαρόζο. Τι, τι θα γίνει με τη Λετωνία, τι θα γίνει ε, με την ε, ανισορροπία που υπάρχει για τις μικρομεσαίες της επιχειρήσεις. Διότι οι πλούσιοι ξένοι αγοράζουν τη γη στη Λετωνία και ε, φυτεύουν ε, και δημιουργούν ε, νέα προγράμματα όπου οι Λετονοί δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας και αναγκάζονται να μετα με κομίσουν στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά ελπίζω να ακούτε αυτά τα οποία ζητούν οι πολίτες μας. Νομίζω τώρα θα επανέλθουμε στον αρχικό ο κατάλογο. Ο κύριος Κανδαλίδης από την Ελλάδα, ο κύριος Υπουργός, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου που ήταν αναγκασμένος να μείνει στην Αθήνα. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνεδρίαση που έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα. Τέτοιες ε, συζητήσεις ε, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να οδηγηθούμε σε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ε, των πολιτών και του αγροτικού κόσμου έχουμε όλοι αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ΚΑΠ. Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζουμε ότι οι προτάσεις της δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές προσδοκίες των Ευρωπαίων αγροτών. Και θα ήθελα να αρχίσω από το θέμα του προϋπολογισμού. Ακροβατούν οι προτάσεις της Επιτροπής μεταξύ φιλόδοξων στόχων και δημοσιονομικών περιορισμών αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία είναι όμως ο μόνος τομέας πολιτικής για τον οποίο προβλέπονται μειώσεις των πόρων. Επίσης δεν συμφωνούμε με τη σύνδεση της δημόσιας στήριξης προς τη γεωργία με τις δημοσιονομικές δυσχέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ε, τέτοιου είδες, είδους ε, ε, ρήτρες οικονομικών κυρώσεων θεωρούμε ότι ακυρώνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. Όσον αφορά την ανακατανομή των συνολικών πόρων, θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί σταδιακά, να υπάρξει μια μεγάλη μεταβατική περίοδος. Για τις άμεσες ενισχύσεις, το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να οδηγεί στην απλούστευση και στην ευελιξία της εφαρμογής ώστε να μην απειλείται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η περιφερειοποίηση των ενισχύσεων είναι ένα μέτρο κοινωνικά δίκαιο. Οφείλει όμως να αντανακλά σε κάθε περιφέρεια τις πραγματικές ανάγκες της γεωργίας με ευέλικτους και σαφείς κανόνες. Το πρασίνισμα της ΚΑΠ θα πρέπει να είναι ένα καθεστώς περιβαλλοντικών κινήτρων. Απλό, κατανοητό και εφαρμόσιμο σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους και σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. Οι υποχρεώσεις για τους γεωργούς θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, ώστε να μην τους αποθερίνουν στην εφαρμογή του πρασινίσματος και να μην τους επιβαρύνουν δυσανάλογα αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ήδη επιφορτισμένοι με αυστηρές απαιτήσεις. Αν ε, τα μέτρα είναι μη ρεαλιστικά, φοβούμαστε ότι θα οδηγηθούμε σε αντίθετα από τα προσδεκόμενα αποτελέσματα, στην αποθάρρυνση των γεωργών να τα εφαρμόσουν. Η καλύτερη στόχευση της δημόσιας στήριξης είναι και αίτημα της κοινωνίας και προϋπόθεση για να διατηρήσουμε το μοντέλο γεωργίας που προωθούμε στην Ευρώπη, τη βιοπικιλότητα, τις πολυλειτουργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται μάλιστα σε συνθήκες λιγότερο ανταγωνιστικές, αλλά που ταυτόχρονα προσφέρουν ουσιαστικά δημόσια αγαθά. Τα όρια που τίθενται για το κάπινγκ θα μπορούσαν να μειωθούν και η προτινόμενη διαχείριση του προϊόντος του κάπινγκ, των πόρων που προκύπτουν, ε, θεωρούμε ότι είναι οπισθοχώρηση σε σχέση με τη σημερινή δυναμική διαφοροποίηση που είναι ένα μέτρο ανάλογης φιλοσοφίας. Από την άλλη πλευρά, ο ορισμός που προτείνεται για τον ενεργό αγρότη θα πρέπει να βελτιωθεί, να δίνει ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να τον αξιοποιούν παραγωγικά και να εκπληρεί το σκοπό του για την αγροτική ανάπτυξη και συγκεκριμένα για την ανακατανομή των πόρων ε, δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο σημερινές ισορροπίες. Στα κριτήρια για την ανακατανομή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που είναι βέβαιο ότι είναι δυσμενέστερες για ορισμένες περιφέρειες της Ένωσης Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου, τα μέτρα για τη σταθεροποίηση των τιμών και των αγορών, καθώς και τα μέτρα για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, είναι απαραίτητα για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη βιωσιμότητα του τομέα, αφού οι κινδυνοί από τις αγορές και τα φυσικά φαινόμενα γίνονται διαρκώς συχνότεροι και εντονότεροι οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν ορισμένα θετικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μπροστά μας μια δύσκολη πορεία μέχρι να φτάσουμε στις τελικές μας αποφάσεις, αλλά από κοινού, με δεδομένη τη βούλησή μας, είναι βέβαιο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε πολιτικές που εγγυώνται ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, αναπληρώτρια του κυρίου Σκανδαλίδη και θα ήθελα να περάσω στην επόμενη ομιλήτρια, η ομιλητή των Σάιμον, Σάιμον Κόνβενι από την Ιρλανδία. Ε, αγαπητοί υπουργοί, κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ε, χαίρομαι για αυτόν τον διάλογο. Είμαι πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από κάποια χρόνια, τώρα υπουργό. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, αυξημένη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αναζήτηση μιας λύσης ε, κοινή αποδοχής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ο διάλογος λοιπόν αυτός αποτελεί την αφετηρία μιας μακράς διαδικασίας που ελπίζω πως θα δώσει ένα αποτέλεσμα αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τη γεωργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνουμε ε, την βιώσιμη εντατικοποίηση ε, της παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα, κάτι που το χρειάζεται και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, αλλά με τρόπο που θα σέβεται τον πλανήτη μας και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η τροφή. Ξέρω ότι είναι περιορισμένο ο χρόνος μου, συνεπώς θα αναφερθώ σε ορισμένες Προτάσει ε, τι οποίε έχει υποβάλει η Κομισιόν θα ήθελα να τι σχολιάσω. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την κατανομή πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί δυσκολίε σε πολλά κράτη-μέλη. Από τη δική μα πλευρά, από την πλευρά τη Ιρλανδία, καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε την ρεαλιστική μέθοδο που προτείνει η Κομισιόν ω ε, βάση για την ανακατανομή. Αλλά με μετεπιτάσεως λέμε πως ε, όταν, παρόλο ότι η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για τον, πυλώνα, τον πρώτο πυλώνα της άμεσης ενισχύσης, δεν είναι σαφές το ποια μέθοδος θα εφαρμοστεί για το δεύτερο πυλώνα. Συνεπώς θα πρέπει η συζήτηση να εξασφαλίσει, ε, να, μάλλον να, θα πρέπει να δούμε πρώτα τη λύση και για το δεύτερο πυλώνα πριν δεχτούμε τη λύση για τον πρώτο. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των κρατών μελών εντό του κάθε κράτους, ε, την πόρων εντό του κάθε κράτου μέλους, αυτό είναι δύσκολο για τη χώρα μου το θέμα. Ε, η, η πρόταση που κάνει ε, η Κομισιόν ανα, η στραματική ενίσχυση μας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Γιατί έχουμε πολλά διαφορετικά συστήματα παραγωγής, έχουμε μια ιστορική υποστήριξη της παραγωγικότητας από τα προηγούμενα συστήματα πληρωμών της ΚΑΠ. Συνεπώς, η, τον, η, απλή και αυτόματη μετάβαση σε ένα ε, στρεματικό σύστημα ε, στο οποίο οι ιδιοκτήτες δεν είναι καν γεωργοί οι αγρότες, θα μας δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα και ενδεχομένως θα πλήξει πάρα πολύ και την παραγωγικότητα και την ε, παραγωγή μας. Ας το σκεφτούμε αυτό και ας επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να έχουν την ευελιξία ε, να επιλέξουν τη λύση που είναι πιο προσαρμοσμένη στη δική τους πραγματικότητα. και ας εξασφαλίσουμε και ότι η Κομισιόν θα έχει ένα σύστημα που θα επιβεβαιώνει πως η λύση που θα επιλέγεται κάθε φορά σε εθνικό επίπεδο δεν θα πλήττει τον ανταγωνισμό, ούτε θα τον αλλοιώνει κλπ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επιλέξουμε ένα μοντέλο ενιαίο για όλα τα κρατημέλη δεδομένη τη ε, ποικιλία περιπτώσεων και καταστάσεων που υπάρχουν στα κρατημέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευελιξία Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων που θα ορίσει η Κομισιόν ή συγκεκριμένων αρχών που θα ορίσει η Κομισιόν και θα αφορούν όλες τις χώρες. Ίδια προσέγγιση και για τα μέτρα πρασινίσματος. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να κάνετε, το υποστηρίζω, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα ηγείται του κόσμου με παραγωγή τροφίμων ε, φιλική προς το περιβάλλον με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και πάλι να έχουμε κοινού κανόνες για όλες τις χώρες. Μια χώρα που είναι στη Μεσόγειο με μια χώρα που βρίσκεται στη Σκανδιναβία ε, έχουν πολύ διαφορετικό κλίμα, ε, πολύ διαφορετικές ποικιλίε, πολύ διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα κλπ. Θα μπορούσατε να υποβάλλεται ένα μενού με δυνατές επιλογές ε, στα κράτη-μέλη και το κάθε κράτος να επιλέξει την, τη δυνατότητα που του ταιριάζει και πάλι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα ελέγχει η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τους νέους γεωργού, συμφωνώ με τις προσπάθειές σας, Επίτροπε, συμφωνώ με την προσέγγιση σα να είναι υποχρεωτικά τα μέτρα αυτά. Θα πρέπει να δραστήρια να ενισχύσουμε τους νέους γεωργούς και να τους υποστηρίξουμε στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Όμως, στην χώρα μου, δυστυχώς, μόνο 7% των γεωργών έχουν ηλικία κάτω από 25 χρόνια. Είναι κάτω των 25 ετών. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια για το πώ θα αναδιανεμηθούν οι πόροι. Αυτό το είπα και προηγουμένω. Όμω ε, έχετε τη σωστή προσέγγιση για το πώ θα δαπανηθούν αυτά τα ποσά. Ε, καινοτομία και ξυγχρονισμό των αγροτικών συστημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο των προτάσεών σα. Ε, υπεύθυνη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, ασφάλεια των τροφίμων, παραγωγικότητα και αποδοτικότητα είναι όλα πολύ σημαντικά και θα βοηθήσουν τους γεωργούς μας να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Τώρα, για την διαχείριση των κρίσεων και την υποστήριξη των ε, αγορών, νομίζω ότι ε, έχετε δίκιο στις προτάσεις σας, ε, είναι αρκετά σωστές. Προτιμάτε να προτείνετε να διατηρήσουμε την παρέμβαση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σε ό,τι αφορά την διαχείριση των κρίσεων. Ελπίζω η Κομισιόν να μπορεί να, απαντά καλύτερα, να αντιδρά πιο γρήγορα σε τροφιμικές κρίσεις όπως ε, δεν έχουμε καταφέρει στο παρελθόν. Είναι πολύ καλό, καλό σημείο κίνηση αυτή η πρόταση. Ε, έχουμε πολλά να κάνουμε το επόμενο εξάμεινο. Συνεπώς ε, ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε τα τρία θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποδεκτό συμβάσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. τώρα τελείωσε θα δώσω μάλλον το λόγο στον κύριο Άγνο και μετά στον κύριο Μαγκίνης, αλλά για τρία λεπτά παρακαλώ να σεβόμαστε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στο πρασίνισμα, σε αυτή την πτυχή του θέματος. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο οι γεωργοί λαμβάνουν ήδη αποφάσεις λόγω αυτών των προτάσεων. Και οι αποφάσεις που λαμβάνουν είναι ζημιογόνες για το περιβάλλον. Αυτοί λοιπόν οι γεωργοί αποφάσισαν να μην συνάψουν περιβαλλοντικές συμβάσεις με το Κοινοβούλιο. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα σύστημα όπου μπορεί κανείς να ενταχθεί σε κάποια περιβαλλοντικά προγράμματα ε, για κάποια χρόνια και υπογράφει κανείς μία σύμβαση. Αυτό για το οποίο ανησυχούν οι Γεωργοί είναι ότι αν συνεχίσετε συμβάσεις για 4-5 χρόνια αυτά θα προστίθενται στο 7% ε, που ε, προβλέπετε εσείς. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ταχύτατα αντιδράσεις, γιατί αν δεν γίνει κάτι, οι γεωργοί αυτοί θα υπογράψουν αυτές τις περιβαλλοντικές συμβάσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι οι βιολογικές καλλιέργειες ε, εξαιρούνται. Γιατί όμως ε, αυτοί οι ε, βιολογικοί καλλιεργητές να έχουν αυτό το προνόμιο έναντι των υπολείπων. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα της συγκομιδής, πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι ε, πολλοί έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή. Όσοι τώρα είναι ε, κάτω από 200 εκτάρια, είναι πολύ ε, πιθανόν την συγκομιδή να την παίρνει ένας ε, διαμεσολαβητής που είναι ένας ε, μεγάλος γεωργός και αυτός και ενδέχεται ο διαμεσολαβητής ε, να επιμείνει όλη η σοδιά να συλλέγεται για ένα χρόνο, του χρόνου άλλη σοδιά ε, και μετά πάλι διαφορετική. Έτσι λοιπόν οι μικροί γεωργοί θα πρέπει σε διάφορες χρονιές ε, να μοιράσουν την παραγωγή τους. Ε, όταν μπαίνουν οι μηχανές δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι καλή η παραγωγικότητα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να δείτε λιγάκι το θέμα του κατοφλιού και να το αυξήσετε σημαντικά μέχρι και 500 εκτάρια, δηλαδή αυτό αφορά μόνο τους πολύ μεγάλους ε, γεωργούς. Μας είπαν ότι αυτά τα μέτρα πρασινίσματος αφορούν την κλιματική αλλαγή, δηλαδή αν το 70% της ε, εκμετάλλευσής μου το εξαιρέσω από παραγωγή, τότε υποτίθεται θα βελτιωθεί ε, το κλίμα στον κόσμο, αλλά δεν είμαι σίγουρη για αυτό, κύριο, που είμαι σίγουρη ότι θα πεινάσουν οι άνθρωποι. Πολλοί ανησυχούν για τη συγχρηματοδότηση, για το 50%. Ε, φαντάζομαι, έχετε συνειδητοποιήσει, οι προλαλήσαντες, ότι υπάρχουν προτάσεις, ε, στην Πορτογαλία τουλάχιστον, να υπάρξει συγχρηματοδότηση και μέχρι το 90%. Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι η γεωργία στις χώρες που θα έχουν την Προεδρία ε, στο μέσο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως η Κύπρος. Πέρσι τον Ιανουάριο πέρασα κάποιες ε, μέρες στην Κύπρο, καλά οργανωμένη χώρα, καλός ο τουρισμός, ε, αλλά είδα σε όλη αυτή την έκταση της Κύπρου μόνο δύο γεωργικές μηχανές. Η Γεωργία, μάλλον η Κύπρος, δεν έχει εξελιγμένη Γεωργία και δεν μπορεί να επηρεάσει, παραδείγματο χάνει τη Γεωργία ε, της, ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απευθυνθώ στον Κύπριο Υπουργό και να με κοιτάξει τα μάτια να μου πει κατά πόσον πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στις δικές μας απαιτήσεις. Επόμενος, Μαγκίνες παρακαλώ. Ε, και άλλη μια έτσι πρόκληση ε, θα επιμείνω στο θέμα των άμεσων πληρωμών. Ε, εδώ και δύο ώρες ε, μιλάμε και η λέξη ευελιξία είναι αυτή που πιο πολύ έχει αναφερθεί από τους υπουργούς και συνεπώς ο Επίτρος θα πρέπει να τη λάβει υπόψη της, να λάβει υπόψη του, να λάβει υπόψη του αυτά τα αιτήματα για ευελιξία. Γιατί είναι αδύνατον το ίδιο καθεστώς να εφαρμοστεί σε όλους. Ε, σίγουρα εμείς που καταλαβαίνουμε από γεωργία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με ένα ενιαίο μοντέλο σύστημα πληρωμών. Ελπίζω ότι στο τέλος της συνεδρίας επίσης θα καταλήξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα ε, για να καταλάβουμε ε, υπό τι πίεση θα λειτουργήσουμε. Καταλαβαίνω ότι ο Επίτροπος ε, ε, θέλει ε, οι προτάσεις αυτές να αρχίσουν να εφαρμόζονται πρώτη 1η του 2014. Ίσως όμως ακούγοντας τις απόψεις σήμερα θα είναι λίγο δύσκολο να προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως μπορούμε να εργαστούμε βάσει αυτή την προθεσμία. Ο κύριος Λαβία μίλησε για το θέμα του προπολογισμού και τα όσα είπε μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα. Συνεπώς, πριν φύγουμε, ίσως θα έπρεπε να δούμε με τους συναδέλφους μας, να πάρουμε μερικά τηλέφωνα για να δούμε πού βρίσκονται οι συζητήσεις για τον περιπολογισμό. Μετά, μην ξεχνάτε το θέμα της πράσινης γραφειοκρατίας. Το έχουμε ξαναπεί, είναι μια έκφραση που λέγεται όλο και περισσότερο τελευταία, διότι πολλά από αυτά τα πρασινίσματα θα οδηγούν σε αύξηση της γραφειοκρατίας. Αυτό το είπαν και πολλοί από τους υπουργούς σήμερα. Δεν φαντάζομαι να θέλετε κάτι τέτοιο. Σίγουρα ούτε και το Κοινοβούλιο θα το επιτρέψει. Γιατί οι γεωργοί συνεχώς μας μιλούν για αυτό το εμπόδιο που είναι η γραφειοκρατία ε, στην καθημερινή ζωή. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για το πρασίνισμα, καταλαβαίνουμε την ανάγκη ε, και καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο σαφής αλλά ε, η υπερβολική λεπτομέρεια δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει να διευρύνουμε λίγο την έννοια του πρασινίσματος. Στη δική μου χώρα υπάρχουν 40 ε, αποχρώσεις του πράσινου. Ε, και νομίζω ότι σίγουρα η Γεωργία θα πρέπει να είναι πιο αυτάρκης σε σχέση με τους πόρους της, να αντιμετωπίζει, να βοηθάει στην αντιμετώπιση του, των, της κλιματικής αλλαγής, των προβλημάτων του περιβάλλοντος κλπ. Αυτές θα πρέπει να είναι οι γενικές αρχές. Αλλά πολλά μέτρα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι προτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακατανομή των πληρωμών, τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και στο εσωτερικό του κάθε κράτου μέλου. Καταλαβαίνουμε πόσο περίπλοκο είναι και ακαθόδε. Δεν θα ήταν πρόβλημα, ε, δεν θα ήταν δύσκολο και ακαθόδε αν ο προπολογισμό δεν δημιουργούσε προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο είπα και προηγουμένω ότι ίσω θα πρέπει να ξέρουμε πρώτα ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα διαθέτουμε. Εν πάση περιπτώσει όμω, ε, στο θέμα τη ανακατανομή θα πρέπει να καταλάβουμε τι συνέπειε. Τόσο στο εσωτερικό του κάθε κράτου μέλου, όσο και στην κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Και θα πρέπει να ακούσουμε όλε τι απόψει. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να καταλήξουμε συμφωνία μεταξύ όλων. Συνεπώς Ευχαριστώ και την Κομισιόν και το Συμβούλιο και εμείς οι ίδιοι θα κάνουμε προσπάθειες ε, επικοδομητικά. Γιατί τελικά κάποιοι μας ακούν, οι οποίοι θα προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους από το 2014 και μετά. Και μας ακούν και οι καταναλωτές που ζητούν και χαμηλές τιμές και καλή ποιότητα. Ταυτόχρονα περιμένει και το περιβάλλον από μας. Συνεπώς είναι πολύ σοβαρός και κρίσιμο ο ρόλο μα. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο σε τρεις ξεκινώντας από τον ε, Ιταλό Υπουργό ε, Γεωργίας ε, και θα ακολουθήσουν δύο συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη διαθεσμική συνάντηση και όντως πρέπει να δημιουργήσουμε από κοινού Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική, η οποία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήση του μέλλοντο. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι οι γεωργοί πρέπει να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί για να μπορούν να ταπεξέλθουν στην παγκόσμια αγορά. Επίση, ε, πρέπει, ζητάνε αυτοί να υπάρχει λιγότερο γραφειοκρατία, πιο απλοί κανόνε. Ε, για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, θα πρέπει την προσοχή μα να την εστιάσουμε στην παραγωγή και στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Και δυστυχώ λυπάμαι, αλλά αυτή η πρόταση της Κομισιόν δεν πάει στη σωστή κατεύθυνση. Η Κομισιόν προτείνει άμεσες ενισχύσεις, πολύ περίπλοκο σύστημα που θα συνεπάγεται ένα βάρος, μεγαλύτερο βάρος για τους γεωργούς. Παράδειγμα, αυτά τα μέτρα για το πρασίνισμα θα είναι επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, δύσκολο να ελεγχθούν και δεν θα προστατεύουν και το περιβάλλον. Επίσης θα είναι ε, και κατά των συμφερόντων της ε, Γεωργίας ε, στην χώρα μου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπάρχουν σωστοί έλεγχοι στα κράτη-μέλη. Είναι άχρηστο να εισάγει κανείς ε, μία λέξη, απλά ένα σλόγγαν, δήθεν για να αποφύγει τα ζυζανιοκτώνα και τα αυτοφάρμακα στην Γεωργία. Κάτι άλλο. Θα πρέπει επίσης, όπως σας είπα, το θέμα των ενισχύσεων είναι θέμα κάθε κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόταση δεν αφήνει στο κράτος μέλος ε, την ευελιξία κυρίως όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις. Και εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όλο αυτό το σχέδιο που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να πλουστευτεί περαιτέρω, ε, να μην υπάρχει βάρος για τις επιχειρήσεις και να ε, δίνει τη δυνατότητα επικουρικότητα στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην αγορά, αυτά θα δοκιμαστούν. Είναι δύσκολα για τους πολίτες. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι η κοινή κυρική πολιτική δεν επιτρέπει στους παραγωγούς να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις ε, αγορές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα για να ε, έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να προσφέρουμε κίνητρα και παράλληλα είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η όλη αλυσίδα, η αλυσίδα παραγωγής και η τροφιμική αλυσίδα. Ε, την επισήμανση των προϊόντων και αυτή οφείλουμε να την προβάλλουμε. Κυρίως ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν προϊόντα από την Αμερική, αμερικανικής προέλευσης, ε, τα οποία δυστυχώς έχουν προνομιούχα μεταχείριση. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα, εκεί πρέπει πράγματι να λάβουμε σημαντικά μέτρα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Και για να τα επιτύχουμε όλα αυτά, δεν μπορούν να ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν τώρα. Η πρόταση Κομισιόν ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση και απομακρύνει διευρύνεται από τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Εγώ λοιπόν θέλω να επισημάνω ότι παραμένει ανεπίλητο το θέμα των πόρων για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν περιφερειακό σχεδιασμό. Τέτοιου είδους χώρε, όπως η Ιταλία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής ευελιξίας και είναι απαράδεκτο ε, κράτη-μέλη τα οποία έχουν περιφερειακή δομή, ε, τα κράτη αυτά να αντιμετωπίζονται όπως και τα άλλα που έχουν συγκεντρωτική μορφή θα πράγματι ε, η κατανομή θα πρέπει να γίνεται και στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα. Εγώ εκείνο που επιθυμώ να υπογραμμίσω είναι ότι η Ιταλία θεωρεί απαράδεκτο λύσεις που θα βρεθούν να μην προβλέπουν ανακατανομή των πόρων κυρίως όσον αφορά την επιφάνεια, τις γεωργικές εκτάσεις. Εμείς επιθυμούμε να λαμβάνεται υπόψη εργασία και πολλοί άλλοι παράγοντες. Ε, γιατί πραγματικά θα ήταν τραγικό αν η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα της παραγωγής θυσιάζονταν μόνο και μόνο για να διατηρηθούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εμείς ως Ιταλία δεν μπορούμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό Γεωργίας της ε, Λετωνίας ε, Λέμντο Στραγιούμα και ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, αν δεν προφέρω σωστά το όνομα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, κύριε Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καταρχήν ε, ε, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την κοινή αυτή συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, η χώρα μου θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής είναι θετική. Αλλά υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να δεχθούμε τη θέση αυτή διότι δεν είναι αποδεκτή για τους γεωργούς μας να έχουν αυτό το επίπεδο αμέσων πληρωμών. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω εδώ μερικούς αριθμούς διότι στην ε, Λετωνία θα έχουμε ε, 1.200 αναεκτάριο ε, ε, ανά εκτάριο και αν το συγκρίνουμε με άλλες χώρες θα δούμε ότι υπάρχει μία τριπλή διαφοροποίηση. Βεβαίως θα μου πείτε ότι είναι διαφορετικό το επίπεδο των πόρων αλλά αν λάβουμε υπόψη την πληρωμή ε, εις μισθούς για το εργατικό δυναμικό θα δείτε ότι οι αριθμοί διαφοροποιούνται και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους γεωργούς μας αυτή τη διαφοροποίηση διότι θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να λαμβάνει κάτι λιγότερο από το 20% του μεσοόρου και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν μόνο έξι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή. Ως εκ τούτου είναι βασικό να υπάρχει διαφάνεια για τις κατανομές στο δεύτερο πληρώνα αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι 5% του δεύτερου πυλώνα πρέπει να κατανεμηθεί ε, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσει τις πληρωμές στον πρώτο πυλώνα και για τη Λετωνία αυτό δεν ε, μπορεί να δημιουργήσει παρά ένα ακόμη πρόβλημα. Εμείς δηλαδή μαχόμεθα υπέρ μια ισότητος εις ε, τις άμεσες πληρωμές και γι αυτό, αυτό χρειαζόμαστε για να συνενέσουμε και τώρα ο Λιθουανός Υπουργός Στάνος ε, ε, Λουκετζεύσκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επιτροπέ κυρίε και κύριοι Υπουργοί και Ευρωβουλευτέ. Ε, ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές ε, της ΚΑΠ κατά εφαρμογή της ε, Συνθήκης Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν οι όροι να είναι ίδιοι για όλους. Η διεύρυνση των λειτουργιών και των στόχων της ε, ΚΑΠ ε, απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση ε, για την περίοδο μετά το 2013, γιατί μας περιμένουν σημαντικές προκλήσεις στο περιβάλλον, η, ασφάλεια, η τροφιμική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Με... Δεν είναι εύκολο με μειωμένη χρηματοδότηση να επιτύχουμε πιο αυστηρούς στόχους. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι δύσκολο να έχουμε την ίδια στρεματική ενίσχυση σε όλη την Ευρώπη, διότι είναι διαφορετικές συνθήκες, κλιματικές, κοινωνικές κλπ. Όμως, για την επόμενη περίοδο θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη προσέγγιση και δίκαιη μεταχείριση όλων των κρατών μελών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Είναι δύσκολο επίση να συμφωνήσουμε με τις μεταβατικές περιόδους που προτείνονται. Εμείς ήδη ε, έχουμε υποφέρει από την ε, μεταβατική περίοδο για 7 χρόνια. Δεν θα ήταν δίκαιο ε, να υποστούμε και μία ακόμα μακρόχρονη μεταβατική περίοδο. Και θα πρέπει να φτάσουμε στην αρχή της επόμενης ε, δημοσιονομικής περίοδου στο μέσο όρο των ε, ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανά στρέμα. Θα ήθελα επίσης να πω το εξής. για άλλα στοιχεία της, ε, του μέλλοντο, του, της μελλοντικής ΚΑΠ. Έχουμε κάποιες ανησυχίε σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα και το υποχρεωτικό ποσοστό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, ευελιξία. Και δεν θα πρέπει να έχουμε ε, οροφές στη χρηματοδότηση για την, το πρασίνισμα πριν εξασφαλίσουμε την αναδιανομή των πόρων. Επίσης, χρειαζόμαστε, ε, χρειαζόμαστε ένα ορισμό για τον ενεργό γεωργό και είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των νέων γεωργών. Όμως, οι προτάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να βελτιωθούν για, τον, για τους, για τους ε, ε, ενεργούς γεωργούς, ενώ οι ενισχύσεις στις μικρές εκμεταλλεύσεις δεν θα πρέπει να είναι κοινωνικές ενισχύσεις και κοινωνικές, ε, κοινωνικά επιδόματα. Ε, θα πρέπει να δίδονται για την συνέχιση της ε, διεξαγωγής της αγροτικής και γεωργικής δραστηριότητας και με συγκεκριμένα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για την αγορά, οι αγορές είναι πολύ ανάστατες για αυτό το λόγο χρειάζονται τέτοιου είδους μέτρα. Ο βασικός, τα βασικά μέτρα ε, θα πρέπει να εγγυώνται τη σταθερότητα, αλλά υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να δεχτούμε. Τι ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Δεν υποστηρίζουμε την ιδέα της κατάργησης των ποσοστώσεων για τη ε, ζάχαρη, για παράδειγμα, από το 2015 και μετά. Ευχαριστώ. Ωραία, τώρα είναι η σειρά των Ευρωβουλευτών, ο κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την καινοτόμο και χρησιμότατη για όλους σημερινή κοινή συνεδρίαση. Επιτρέψτε μου δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Στο περίφημο πρασίνισμα φαντάζομαι ότι θα ήταν αποτελεσματικότερο αν παίρναμε υπόψη μας τις ιδιομορφίες και διαφορετικότητες που διακρίνουν τις περιοχές της Ένωσης. Επί παραδείγματι, οι παραδοσιακοί ελαιώνες χαμηλών ισρώων είναι κυρίως ξηρικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούν ελάχιστα φυτοφάρμακα και βελτιωτικά, διατηρούν το παραδοσιακό τοπίο και την πολιτισμική παράδοση, ενισχύουν τη βιοπικιλότητα, συντηρούν κοινότητες σε περιθωριακές περιοχές με ελάχιστες επιλογές σε εναλλακτικέ οικονομικές δραστηριότητες και συμβάλλουν στην αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος. Επομένως, καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή. Γιατί λοιπόν οι παραδοσιακοί ελαιώνες όπως και άλλες δενδρώτες καλλιέργειες να μην συμπεριλαμβάνονται στην πράσινη ενίσχυση της νέας ΚΑΠ. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην κρισιμότητα που έχει το θέμα της κατανομής των δημοσιονομικών πόρων για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών και ιδιαίτερα βεβαίως στη σημερινή ιδιαίτερως δύσκολη για όλους συγκυρία είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που θέτει η οικονομική κρίση, ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη-μέλη, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων της ανάπτυξης της υπαίθρου και να αρθεί η απειλή που συνδέει την παροχή στήριξης με τις δημοσιονομικές δυσχέρειες στην Ένωση ή στις χώρες μέλη. Θεωρούμε κρίσιμη επίσης στην επιλογή κριτηρίων για την κατανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα αλλά και για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού έκτακτης ανάγκης την αναγνώριση της επιπρόσθετης επιβάρυνσης που θα υποστεί κατά κοινή ομολογία η γεωργία των χωρών του Νότου από την κλιματική αλλαγή. Θα ήταν τέλος κοινότυπο να προσθέσω πως τα μέτρα για την σταθεροποίηση τιμών και αγορών, τη διαφάνεια των αγορών, όπως και την απλοποίηση, την απογραφειοκρατικοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής ενδιαφέρουν το σύνολο των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων και γεωργών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σπύρο και τώρα έχουμε άλλους τρεις υπουργούς και ξεκινούμε με τον ε, κύριο Σνάιντερ από το Λουξεμβούργο και μετά θα δώσω το λόγο στο Jim Μπέις για το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά τον Σλότ Σάιμον της Σλοβακίας. Ε, κύριε Σνάιντερ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Πάολο Μάρεκ και ε, τον Ντάτσιαν για την σημερινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να προσαρμοστεί η, η γεωργία εις τις προκλήσεις και η διατροφική ασφάλεια πρέπει να είναι ο βασικός στόχος της πολιτικής μας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα ε, προϋπολογισμό που να βρίσκεται στο ύψος των προσδοκιών μας και θα πρέπει να ε, ε, συμπεριληφθεί ο προπολογισμό και του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα για να υπάρχει μία δίκαιη κατανομή. Ε, προσφερόμαστε όπως και στο παρελθόν για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία αλλά έχω ορισμένε παρατηρήσεις. Όσον αφορά τις πληρωμές πρέπει να υπενθυμίσω ότι για το Λουξεμβούργο η αιτιολόγηση των αμέσων πληρωμών αποβαίνει ε, προς όφερος ε, των ε, παραγωγών και για την βελτίωση των κοινών αγαθών που προσφέρει η γεωργία. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα νομίζουμε ότι δεν χρειάζονται περισσότερα περιβαλλοντολογικά κριτήρια ή στις άμεσες πληρωμές διότι η βελτίωση της αναπτύξεως της υπαίθρου είναι πρωταρχική και πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα για να μπορέσουν δε οι με σεγές να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίσουν τη διατροφική ασφάλεια. Όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τους μικρούς παραγωγούς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι θελοντικό. Πολλές πολλές προτάσεις της Επιτροπής θα αυξήσουν τα διοικητικά έξοδα των επιχειρήσεων και των εθνικών διοικήσεων όπως η διεύρυνση της πολλαπλής συμμόρφωσης σε νέους τομείς, η οικολογική πληρωμή και ε, ο καθορισμός του ενεργού γεωργού. Θεωρούμε όμως ότι τα μέτρα γενικώ βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα επιτρέψουν κάποιες κάποια συνέχεια και συνεκτικότητα με τις προηγούμενες περιόδους παρόλο που δεν προβλέπεται μείωση της γραφειοκρατίας για να επιταχυνθεί η αποδοχή των προγραμμάτων, το monitoring και η αξιολόγηση. Η ιδέα της ε, κοινής, του κοινού προγραμματισμού με άλλα προγράμματα και η καινοτομία δεν απλοποιεί τις διαδικασίες χωρίς όμως να προσφέρει και μία προστιθέμενη αξία ιδίως στις χώρες που έχουν μικρά προγράμματα. Τέλος πρέπει να τονίσω την ευαισθησία του θέματος του καθορισμού των μειονεκτικών περιοχών διότι πιστεύουμε ότι ο κατάλογος των κριτηρίων που προτίθεται δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Τέλος, όσον αφορά την διαχείριση των αγορών, στηρίζουμε την ιδέα να υποστηριχθεί η ατομική και ιδιωτική αποθήκευση για να βελτιωθεί το σύστημα και θα πρέπει να υπάρξει μία επέκταση της φυτεύσεως και τέλος λυπούμεθα ότι δεν υπάρχει μία πρόταση για την ομαλή προσγείωση όλων των κρατών ή σε την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων το 2015. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ. Ο κύριος Jim Paynes από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ ε, όλους ε, όσοι συνέβαλαν στο να ε, οργανωθεί η σημερινή συζήτηση. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις για όσο χρόνο χρειαστεί, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια κοινή γεωρική πολιτική που θα είναι κατάλληλη για το μέλλον. Υπάρχουν πολλά τμήματα της πρώτης Κομισιόν που χαιρετίζουμε, την ευελιξία στον δεύτερο πυλώνα και τη δέσμευση της ε, Κομισιόν σε έρευνα και ανάπτυξη και συναφή μέτρα. Από τη στιγμή που ο Επίτροπος έχει κάνει πάρα πολύ για να αυξηθεί η παραγωγή τα επόμενα αιτία, ε, δεν νομίζω ότι αυτό εκφράζεται στις προτάσεις που κατατέθηκαν. Και μάλιστα δεν βλέπουμε τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία δύο-τρία χρόνια όταν οι τιμές των βασικών προϊόντων αυξήθηκαν, οι περισσότερες, των περισσότερων μάλιστα. Και επειδή αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση, ε, βλέπουμε ότι οι τιμές των ε, βασικών αγαθών ε, θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η τάση είναι ανωδική. Πιστεύω λοιπόν ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει αυτά να τα αντικατοπτρίζει και να μην μιλάμε μόνο για το πόσα χρήματα δαπανώνται, αλλά πού ακριβώς δαπανώνται για να λαμβάνεται υπόψη μεταβαλλόμενη κατάσταση. Εδώ λοιπόν χάνεται μια ευκαιρία. Αντί να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα τα κονδύλια για να βοηθηθούν οι γεωργοί της έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αυξανόμενες τιμές ε, που έρχονται λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, ε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στον δεύτερο πυλώνα ως ο, μηχανισμός ε, για να γίνουν οι γεωργοί πιο καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι ο σωστός τρόπος για να ενθαρρύνουμε το πρασίνισμα της ΚΑΠ. Εμείς ε, το κάνουμε αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και αρκετά έτη. Τελικά, αν θέλουμε όμως να έχουμε και πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα, αυτό ε, πρέπει να έχει αξία για τον ε, φορολογούμενο. Επίσης, όλα αυτά πρέπει να είναι απλά. Παραδείγματο χάρη, ο Επίτροπος κατέστησε σαφές ότι το 7% δεν θα αφορά την αγρανάπαυση. Δεν θέλει να εισάγει την αγρανάπαυση. Ε, διότι αυτό είναι θετικό κατά την άποψή μας. Πάντως ε, πολλοί γεωργοί ε, δεν θα έχουν ένα 7% της γης τους που να μπορούν να το αφήσουν σε μη καλλιεργήσιμη έκταση. Ίσως μερικοί να έχουν, αλλά άλλοι πάλι όχι. Και δεν ξέρω τελικά αυτό το 7% πώς θα μπορούν να το βρουν αν δεν αφαιρεθεί γη από καλλιέργειες. Επίσης ε, και άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για το περίφημο κάπινγκ. Ε, νομίζω ότι η διαδικασία ακολουθεί τη λάθος κατεύθυνση. Έχοντας ακούσει τους υπουργούς και συναντέλφους από τη Γεωργική Επιτροπή, εγώ καταλήγω στο ότι η έννοια της σύγκλησης των πληρωμών σε ένα κράτος μέλος δεν είναι αποδεκτή και ελπίζω η Κομισιό να αποσύρει αυτή την πρότασή της. Στηρίζω όλα αυτά που λέχθησαν σήμερα σχετικά με την απλούστευση. Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό. Είναι ένας ευγενής στόχος, αλλά δεν πιστεύουμε ότι οι προτάσεις όσες έχουν τώρα μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Ε, τώρα ο Σόλτ Σάιμον, ε, Υπουργό Γεωργίας της Σλοβακίας. Καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου για αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι πολύ συχνό οι υπουργοί να βρίσκονται και να συζητούν εδώ, στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκ μέρου της θέλω να πω ότι οι προτάσει ε, μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ ήταν μια σχετική απογοήτευση για μας. Δεν είναι επαρκής ε, για να, αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστούν οι, οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δίδεται η υπερβολικά πολύ έμφαση στο πρασίνισμα κάτι που θα μας δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στο μέλλον. Συνεπώς, ε, έχουμε επιφυλάξεις για μια σειρά στοιχείων των προτάσεων της Κομισιόν. Καταρχήν, να μιλήσω για το γεγονός ότι χρειαζόμαστε ίδιους κανόνες για όλους στην εσωτερική αγορά, στην ενιαία αγορά. Πώς είναι δυνατόν να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο όταν ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή έχουμε διαφορετικές ενισχύσεις για το ίδιο αγαθό. άλλες ενισχύσεις να πληρώνονται στη Δανία και άλλες στη Λιθουανία για, το, για την ίδια παραγωγή. Θα πρέπει αυτές οι ενισχύσεις να συγκλίνουν. Νομίζουμε ότι η μεταβατική περίοδος των 7 ετών για τα νέα κράτη-μέλη είναι επαρκής περίοδος, ήταν επαρκής περίοδος, δεν χρειαζόμαστε άλλη μεταβατική περίοδο. Το 30% των πόρων για το πρασίνισμα με 7% εγκατάλειψη γεών θεωρούμε ότι δεν είναι προτάσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγής. Αντιθέτως, θα οδηγήσουν στη μείωση της παραγωγής. Το 30% των πόρων στην, ε, στο πρασίνισμα θα δημιουργήσει, θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Όχι σε αύξηση της παραγωγής. Θα πρέπει το ποσοστό αυτό να μειωθεί. Και ε, μάλιστα να γίνει και εθελοντικό, όχι υποχρεωτικό. Σε ό,τι αφορά το κάπινγκ, τις οροφές, ε, διαφωνούμε με αυτές τις προτάσεις. Ελπίζουμε ότι ο Επίτροπος θα τις αναθεωρήσει και δεν θα τις, εφαρμόσει. Δηλαδή, ε, οροφές στις ενισχύσεις ε, δεν οδηγούν σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο ορισμός του ενεργού γεωργού είναι καλοδεχούμενος αλλά το 5% δεν είναι επαρκές. Το ποσοστό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 30%. 30% του εισοδήματος του συγκεκριμένου να προέρχεται από τη Γεωργία. Ε, η κατάργηση των υποσυστημάτων πληρωμών επίσης δεν είναι ε, απλοποίηση. Πώς είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε τους γεωργούς όταν τους νέους γεωργούς όταν το 2014 κανένας δεν θα είναι δικαιούχος να λάβει ενίσχυση δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθεί ως, ιστορική, ως αναφορά ιστορικά ε, το 2011. Ε, ε, αν θεωρήσουμε ως ε, έτος αναφοράς του 2011 δεν θα υπάρχουν και νέοι γεωργοί ούτε μικρές εκμεταλλεύσεις στο μέλλον. Καινούριες μικρές εκμεταλλεύσεις. Μετά για την ε, κατάργηση των ποσοστώσεων της ζάχαρης το 2015. Στο Συμβούλιο είχαμε πει ότι οι αποφάσεις που, είχαν, που, που ελήφθησαν θα είχαν αρνητικές επιδράσεις και το είδαμε τελικά. Γι' αυτό το λόγο διαφωνούμε την ε, πρόταση της Κομισιόν. Τώρα λοιπόν ε, περνάμε πάλι στους ε, βουλευτές. Ο Αντιπρόεδρος Πόλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους υπουργούς και όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ. Σας δίνω λίγα λεπτά για να μπορέσετε να βάλετε τα ακουστικά σας. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής, πρέπει να πω ότι ε, περιέχει πολλές, πολύ καλές προτάσεις. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα του να τονιστού στη ο ρόλος των γυναικών και μάλιστα των νέων γυναικών που θέλουν να παραμείνουν στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι οποίες δυσκολεύονται να εξασκήσουν γεωργικά επαγγέλματα και μιλάμε για οικολογία, για ένα συμπαθητικό φυσικό περιβάλλον γιατί λοιπόν να μην καθορίσουμε σαν ρεαλιστικό στόχο, εάν θέλετε, να μπορέσει η γεωργία και η δασοκομεία να γίνουν αυτάρκης μακροπρόθεσμα και να δημιουργήσουν ενέργεια για την Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη ε, έχουμε τα περιτώματα των ζώων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενέργεια. Ε, βέβαια ε, Υπάρχουν προβλήματα, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο κύριε Επίτροπε. Ξέρετε ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε ε, τα ε, ορυκτά καύσιμα και πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις ε, για να υπάρχει πιο οικολογική πτυχή. Αντιλαμβάνομαι ότι τα νέα μέτρα είναι πιο γραφειοκρατικά από ό,τι πράσινα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια επιδότηση ε, για τη διαφορά των τιμών μέχρι την αγορά. Αυτό όμως τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει με τρόπο πολύ πιο απλό, πιο άμεσο θα πρέπει οι γεωργοί να ανταμείβονται ε, για τις ε, πολιτιστικές και οικολογικές προσπάθειές τους, διότι αυτοί παράγουν και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα οι δύο τελευταίοι υπουργοί. Δίνω τον ε, λόγο στον Γιάρη Κώστιανεν, υπουργό της ε, της Φιλανδίας και θα ακολουθήσει ο Ρουμάνος Υπουργός. Ευχαριστώ. Ε, Επίτροπε, Υπουργοί, μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ για την οργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Είναι μια πολύ καλή αφετηρία για την συνεργασία μεταξύ των τριών οργάνων. Θέλω να σχολιάσω τα εξής, να υπογραμμίσω τα εξής ζητήματα. Οι νομοθετικές προτάσεις κομισιών θεωρούμε ότι αποτελούν ορθή βάση για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. οι τρεις βασικές ε, αρχές που διέπουν τις προτάσεις Κομισιόν μας βρίσκουν σύμφωνους. Η γεωργία θα πρέπει να γίνει βιώσιμη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι στόχοι που έχει θέσει η Κομισιόν όμως μπορεί να επιτευχθούν με πιο απλό τρόπο. Το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι πολύ περίπλοκο στον έλεγχό του, στη διαχείρισή του και στη λειτουργία του. Η Κομισιόν θα έπρεπε να δώσει περισσότερη έμφαση στην απλοποίηση του συστήματος. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, συμφωνώ με τις προτάσεις της Κομισιόν για τη σταδιακή εξίσωση. Επίσης, συμφωνώ με την διατήρηση των άμεσων πληρωμών. Οι προτάσεις της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικές εκεί που το κόστος παραγωγής είναι ψηλό. Επίσης μας βρίσκουν σύμφωνες οι προτάσεις Κομισιόν για το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα. Όμως θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά τις προτάσεις αυτές για να μην αυξηθεί η γραφειοκρατία. Τρίτον, Δεδομένων των συνδικών που επικρατούν στη Φιλανδία, χαιρόμαστε για τις προτάσεις Κομισιόν για ένα ε, ε, ευρύ πακέτο ε, μέτρων ανάπτυξη πέθρου. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την αγορά, η Κομισιόν έχει δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση των κρίσεων, αλλά η κατάργηση των ποσοστών ζάχαρης με το 2015 δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, εμείς πιστεύουμε ότι η σημερινή συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εδώ συζητούνται προβλήματα ενός κλάδου που είναι πολύ σημαντικός ε, στην Ευρώπη σήμερα και θα είναι και στο μέλλον. Ε, με την πρώτη ματιά τα προβλήματα ναι μεν μοιάζουν είναι πολύ περίπλοκα ε, και είναι πραγματικά επίτευγμα της Κομισιόν το ότι μας καταθέτει αυτές τις προτάσεις. Γιατί οι προτάσεις είναι σημαντικές για το χρονικό διάστημα ε, μέχρι το 2020. Η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική γιατί ε, προλυαίνει το έδαφος ε, για λύση, λύση με πολλές προεκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει η ιδιαιτερότητα των γεωργικών συστημάτων, τι σημαίνει ιδιαιτερότητα της γεωργίας σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ε, ποιες είναι οι απαιτήσει ε, στο εγγύς και στο απότερο μέλλον για την παραγωγή των τροφίμων. Το θέμα δεν είναι να ασχοληθούμε μόνο με την παραγωγή τροφίμων και την εκμετάλλευση των πρώτων υλών. Αυτό που ενδιαφέρει επίση είναι να προσφέρουμε και πρώτε ύλε για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στο μέλλον. Επίση είναι σημαντικό η γεωργία να παραμείνει ποιοτική και ποσοτικά και ποιοτικά και να ε, διαφυλάσσεται η ευθύνη για το εισόδημα των γεωργών και για εκείνους που διαχειρίζονται ένα μεγάλο πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι τα δάση και οι πρώτες ύλε. Επίσης φέρουμε ευθύνη και απέναντι στους ε, καταναλωτές. Εμείς η παραγωγή των ε, τροφίμων ε, φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Εμείς επιθυμούμε να τοποθετηθούμε σε ορισμένα μέτρα όπου πρέπει να υπάρξει αντιλεχής έλεγχος. Πρώτον, πώς θα γίνει η ισότιμη και η ισόποση ε, κατανομή των ε, άμεσων ενισχύσεων. Γιατί υπάρχουν ε, διαφορές στην εκταμείευση κονδυλίων. Σε κάποια κράτη δεν επαρκούν τα κονδύλια. Εξάλλου, στις άμεσες ενισχύσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση της οικολογικοποίησης, όπως λέγεται. Εξάλλου πρέπει να ελέγξουμε και το μήπως αυξάνεται ε, ο κίνδυνος της ε, γραφειοκρατίας γιατί αυτή μπορεί να επηρεάσει τις ε, αποτελεσματικές επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν κατά πολύ στην ασφάλεια τροφίμων και λειτουργούν με υψηλά κριτήρια, με υψηλές προδιαγραφές. αν καταργήσουμε τις επιδοτήσεις ε, επενδύσεων για ορισμένους κλάδους, τότε πλέον θα είναι δύσκολο να έχουμε παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Δυστυχώς τα μέτρα που προτείνονται τώρα δεν είναι ελκυστικά. Αυτά που προτείνονται για τους μικρούς γεωργούς τα χαιρετίζουμε, αλλά πρέπει να δούμε πώς ε, θα οριστεί το ανώτατο ε, πλαφόν. 5.000 ε, αντί για 1.000 ευρώ για τους γεωργούς ε, που δεν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευσή τους ε, και εφαρμόζουν καινοτόμα μέτρα. Πρέπει να συζητήσουμε και για το ποσοστό που αφορά τους νέους γεωργούς. 2% από τον εθνικό προϋπολογισμό και να ισχύει και ένα ποσοστό σε συνάρτηση της έκτασης για την κοινή οργάνωση αγοράς. Πρέπει να επαναφέρουμε τις ενισχύσεις επιδοτήσεων για εξαγωγές, κυρίως για βόλιο κρέας, ε, κρέας ε, χείρων Επίσης, ε, θεωρούμε όσον αφορά την ποσόστοση της ε, ζάχαρης. Εδώ η Κομισιόν πρέπει να αναλύσει ε, τι θα γίνει στην αγορά όταν θα εκπνεύσει η ποσόστοση αυτή το 2015. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει παράταση μέχρι το 2018. Επίσης είμαστε και υπέρ μιας σταδιακής αιτήσιας αύξησης της ποσόστοσης κατά 5%. Αυτό μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις αν υπάρξει κατάργηση της ποσόστοσης. Όσον αφορά τη μελισσοκομεία, εμείς πιστεύουμε ότι εκεί χρειάζονται νέα μέτρα έτσι ώστε να ε, διαδοθεί ε, το μέλι στα σχολεία. Για το γάλα. Εμείς η Ρουμανία πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν καινούργια νέα μέτρα ε, κυρίως ε, όσον αφορά την σύναψη συμβάσεων. Οι συμβάσεις πρέπει να είναι δεσμευτικές. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ ασφαλείας όσον αφορά στο κρέας. Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις στρεβλώση αγοράς για την ανάπτυξη της υπέτρου. Ε, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να αποκλειστούν. Να αποκλείονται οι επιχειρήσεις. Ε, διακόπτεται όμως ο μιλητής. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε λοιπόν με τις παρεμβάσεις των Υπουργών. Βεβαίως είναι σαφές ότι θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στους εκπροσώπους των Υπουργών που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Αλλά μην ξεχνάτε θα είσαστε σύντομοι γιατί έχουμε μόνο 25 λεπτά. Και τώρα όμως θα περάσουμε στους ε, βουλευτές πρώτα. Ε, Όλγα σε σένα είναι ο λόγος. Ευχαριστώ. <clears throat> Σχετικά με την ΚΑΠ όλοι συμφωνούμε με τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα τις κρίσεις, να είναι πιο πράσινη ε, και απλούστερη. Θέλουμε να την ε, ε, ορθολογήσουμε και γι' αυτό πρέπει τώρα να εξετάσουμε μία συγκεκριμένη πρόταση που διατήρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, τα, οι ε, τα διάφορα κράτη έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές απόψεις και αυτό με ανησυχεί. Γιατί αν στην αίθουσα αυτή μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ε, του συνεταιρισμού των γεωργών, ε, δεν μπορέσουμε να προτείνουμε μία νέα κοινή γεωργική πολιτική την οποία να, να προωθήσουμε στους ε, γεωργούς τότε θα είναι εις βάρος όλων μας και οι καταναλωτές και οι ε, γεωργοί θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον σοβαρά προβλήματα γι' αυτό και σας παρακαλώ να είσαστε πιο ανοιχτοί σε συμβιβασμούς για να μπορέσουμε να βρούμε τη σωστή μορφή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αν αυτό δεν γίνει, τότε η ιστορία θα επαναληφθεί. Όπως στην περίπτωση του προϋπολογισμού για να βοηθήσουμε τους φτωχότερους διότι όλοι ήταν υπέρ της προτάσεως αυτής αλλά χάσαμε την μάχη εις ε, την ψηφοφορία. Ωραία. Η Edit Klauser για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι παριστάμενοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην κοινή αυτή ε, συνεδρίαση για να συζητήσουμε την ε, ε, μελλοντική γεωργική πολιτική. Η Αυστρία θεωρεί ότι είναι μία καλή πρότηση αλλά θα χρειαστούν ορισμένες προσαρμογές για να είναι ακόμη καλύτερη και θα βασιστώ και θα περιοριστώ σε λίγες παρατηρήσεις. Καταρχήν τις άμεσες πληρωμές οι οποίες σύμφωνα με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξουν άρδιν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για πολλά κράτη-μέλη και την Αυστρία θα χρειαστεί μία προσαρμογή. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την Αυστρία, την απλοποίηση. Ε, είναι ανάγκη να απλοποιήσουμε και αυτό το τόνισαν πολλές αντιπροσωπές και η Αυστρία ζητά μία πραγματική απλοποίηση της ε, διοικήσεως διότι οι άμεσες πληρωμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν εξετάσουμε τα, τις διάφορες πρημοδοτήσεις αποδεικνύουν ότι το θέμα περιπλέκεται και χρειάζεται ένα πιο απλό σύστημα που θα καταλήγει στον ίδιο στόχο και αναφέρω ένα παράδειγμα παραδείγματος χάρη ε, το ε, την οικολογική πρημοδότηση η οποία όμως περιπλέκει το σύστημα μέσων πληρωμών και θα πρέπει να υπάρξει μία μοναδική πρημοδότηση που θα συγχωνεύει όλες τις προηγούμενες και αυτό αναφέρεται και στην πολλαπλή συμμόρφωση για να περιλάβουμε την οικολογική πτυχή στις εξετάσεις μας. Όσον αφορά την ευελιξία των κρατών μελών πρέπει να υπάρχει για το περιφερειακό πρότυπο, πράγμα το οποίο τόνισαν διάφορες χώρες. Στην Αυστρία έχουμε μια πολυσχηδή γεωργία με πολλές περιοχές και διάφορα είδη πριμοδοτήσεων θα δημιουργούσαν σύγχυση στη χώρα μας και γι' αυτό ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του προτύπου. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου στο δεύτερο πυλώνα είναι πολύ βασικό για μας ιδίω με, το με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και θέλει η χώρα μου να συνεχίσει μία επικερδή ε, εξάσκηση της γεωργίας η οποία όμως χρειάζεται στο σωστό πλαίσιο και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διάφορα πρότυπα και γι' αυτό για την ανάπτυξη της υπαίθρου δεν χρειαζόμαστε επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Για την κοινή διάταξη της αγοράς οι προτάσεις είναι καλές, βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά λιγότερο θετικό είναι ε, η εκπνοή των ποσοστώσεων της Ζαχάρεως και τα θέματα που συμπαρασύρει. Γι' αυτό και ζητούμε να συνεχιστεί αυτή η πρημοδότηση. Τέλος, Όσον αφορά τους άλλους τομείς της γεωργίας υπάρχει ένα κεντρικό θέμα ε, το οποίο απασχολεί και τη χώρα μου και θα εξασκήσουμε μία ε, επικοδομητική πολιτική. Πολύ ωραία. Τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεδομένου ότι δεν έχω και πολύ χρόνο, θα πάω κατευθείαν στην ουσία το πακέτο αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διαπραγματευτική βάση. Μπορεί όμως να βελτιωθεί πολύ, χρειάζεται να βελτιωθεί πολύ. Θα πρέπει να απλοποιηθεί, να δοθεί ε, περισσότερη ευελιξία στο σύστημα ε, και να τονιστεί η επικορικότητα. Για τις άμεσες πληρωμές εμείς υποστηρίζουμε το σύστημα της ανακατανομής ε, των πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη σταδιακή ε, και δίκαιη λαμβάνοντα υπόψη και του δημοσιονομικού προπολογισμού. Ε, πρέπει να εγκαταλείψουμε τι ιστορικέ αναφορέ ε, και να συγκλίνουμε τι ενισχύσει και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Ε, αλλά θα πρέπει το σύστημα να δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, μεγαλύτερη επικουρικότητα, γιατί μέσα στο κράτος, σε κάθε κράτο μέλο υπάρχουν πολλέ πραγματικότητε, οι προτάσει Κομισιόν δεν μα ικανοποιούν. Το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα το έχουμε υποστηρίξει από την αρχή, εμείς ως Γαλλία. Βέβαια, τα συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα δεν μας ικανοποιούν αυτή τη στιγμή, πολύ γραφειοκρατικά, ε, περιτά γραφειοκρατικά ε, και δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικότητες εκμεταλλεύσεις. Η Γαλλία χαιρετίζει την, δυνατότη, την διατήρηση της δυνατότητας ε, ε πληρωμών ε, που δεν θα είναι από συνδεδεμένων πληρωμών από το 2014 και μετά. Ε, επίσης, στη διαχείριση των κρίσεων ε, και, στη διαχείριση των αγορών πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ε, πιστεύουμε ότι τα μέτρα της Κομισιόν είναι θετικά, ε, μπορούν να βελτιωθούν όμως. Για δύο συγκεκριμένα σημεία έχω να κάνω τα εξή σχόλια. Θα πρέπει να εργαστούμε πιο πολύ. Πρώτον, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, δεν μας ικανοποιεί. Δεν θα επιτρέψει την ενίσχυση της συλλογική οργάνωσης ε, των παραγωγών. Θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ στις διαπραγματεύσεις. Δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω το γεγονό ότι στον τομέα τη ζάχαρη η Γαλλία δεν μπορεί να δεχτεί την κατάργηση των ποσοστώσεων του 2015. Επιθυμούμε τη διατήρηση του συστήματο μέχρι το 2020. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα. Ε, οι προτάσει τη ε, Κομισιόν είναι πολύ περίπλοκε, ε, παρόλο που υποτίθεται ότι έχουν ω στόχο την ε, ομογενοποίηση του συστήματο. Εμεί θέλουμε πραγματική πρόοδο, γρήγορη πρόοδο στα, στο θέμα των μειονεκτουσών περιοχών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, το χρηματοοικονομικό κανονισμό διαχείριση τη ΚΑΠ, θα επιμείνω και εγώ στο εξή. Η απουσία πραγματικής απλοποίηση αντίθετα με τα όσα είχε ε, ανακοινώσει η Κομισιόν, ε, δεν μας ικανοποιεί. Τέλος, όλα όσα συζητούμε έχουν νόημα μόνον αν η ΚΑΠ διαθέτει ένα επαρκή ικανοποιητικό προπολογισμό. Αυτό που προτείνεται σήμερα από την Κομισιόν αποτελεί για μας το απόλυτο ελάχιστο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν ο, η εκπρόσωπος της ε, Εστονίας, η Κάτριν Πουν. Παρακαλώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή την ε, πρώτη ιστορική θα έλεγα συνάντηση. Εκ μέρους λοιπόν ε, του Υπουργού Γεωργίας της Εστονίας θα ήθελα να υποστηρίξω δύο θέματα. Για την Εστονία το σημαντικότερο στη συζήτηση ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, είναι οι άμεσες ε, πληρωμές. Η Εστονία στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το επίπεδο των άμεσων ισχύσεων, αλλά δεν συμφωνούμε με το χρονοδιάγραμμα γιατί δεν εγγυάται ε, ίσες ε, προϋποθέσεις για όλους. Εμείς θεωρούμε το δικό μας το επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 90% του μέσου επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι η υποστήριξη της γεωργίας θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο στον επόμενο προπολογισμό και οι άμεσες ενισχύσεις δεν πρέπει να συσχετίζονται με την ανάπτυξη της γεωργίας γιατί αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τις διαρθρωτικές επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να προκύψει ε, ανανέωση και εξυγχρονισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρίως ε, που ήσασταν σύντομοι πρέπει να επιταχύνουμε λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κόστιγκια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι πεπισμένη ότι η ασφάλεια, η τροφιμική ασφάλεια ε, πρέπει να προβληθεί περισσότερο, γιατί έχει σχέση με τους ε, καταναλωτές. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μας μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις της ε, Κομισιόν όσον αφορά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και τις ε, οικολογικές πρημοδοτήσεις. Βεβαίως δεν καλούμεθα <clears throat> να επανανακαλύψουμε τον τρόχο, αλλά να δούμε τι λειτουργήσε σωστά και τι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Από την επανάσταση να περάσουμε στην εξέλιξη. Ε, το 5% της αγρανάπευσης, αυτό που προτάθηκε, θα οδηγήσει σε επανάσταση, κυρίως ε, στις τάξεις των ε, γεωργών και αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία μέτρα έτσι κι αλλιώς ελήφθησαν πολλά μέτρα όπως ο αναδασμός Αυτά τα 10% τελικά όμως αφαιρέθηκαν από τους γεωργούς. Ε, όπως και οι προηγούμενοι και οι προαλήσαντες και εγώ ε, είμαι πολύ επιφυλακτική όσον αφορά την ε, γραφειοκρατία που θα αυξηθεί αν τελικά υπάρξει το πρασίνισμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ε, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι άμεσες ενισχύσεις ε, των γεωργών. Εδώ πρόκειται για την πολλαπλή συμμόρφωση και θεωρώ ότι είναι δικό μας ε, καθήκον να ενημερώσουμε καλύτερα τους άμεσα ενδιαφερόμενους στην κοινή γεωργική πολιτική. Ας μην ξεχνάτε ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι η αξιοπιστία και απέναντι στους ε, καταναλωτές και απέναντι στους ε, γεωργούς, γιατί αυτοί εργάζονται σε καθημερινή βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση που θα είναι συνεργασία ανάμεσα στους γεωργούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε σωστούς κανόνες που θα είναι εύκολο να τηρηθούν επίσης ενδιαφέρει είναι ότι το ε, πρασίνισμα αποδυναμώνει το δεύτερο πυλώνα που είναι όμως η καρδιά της ε, γεωργικής πολιτικής. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε τα κράτη τα οποία την τελευταία δεκαετία προσέφεραν τόσα πολλά να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Πολλά σημεία από αυτά που πρότεινε ο Επίτροπος τα βρίσκω πολύ σωστά, κυρίως την τόνωση της ε, καινοτομίας, το θάρρος ε, για επενδύσεις και επίσης ε, και το ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα ως προς την ασφάλεια των πρώτων υλών. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Το να εκπνεύσει η ποσόστοση ζάχαρης το 2015 δεν είναι και πολύ σωστό. Στη βιοενέργεια και εκεί πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα. Και είμαι αισιόδοξη ότι από κοινού όλοι μαζί θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κόστιγκερ. Τώρα έχουμε την εκπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο, ε, τον εκπρόσωπο της ε, Ουγγρικής ε, Γεωργίας. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη της Ουγγαρίας θα χρειαστούμε μία ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική για το μέλλον της Ευρώπης με ευρεία στήριξη τουλάχιστον ε, εισάξια του παρελθόντος και ναι μεν έχουμε μία καλή βάση διαπραγματεύσεων αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να βελτιώσουμε το κείμενο. Η Ουγγαρία πιστεύει ότι στο μέλλον θα πρέπει να παράγουμε τρόφιμα με τρόφιμα τρόπο ανταγωνιστικό και αν, το αν θα κρατήσουμε τους δύο πυλώνες της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι κάτι συμπεφωνημένο αφενός για το σταθερό εισόδημα των γεωργών αλλά και για να έχουν ευελιξία τα κράτη-μέλη για το πώς θα χρησιμοποιήσουν την στήριξη αυτή. Το κατόφλι του 10% είναι θετικό για τις ευαίσθητες περιοχές εμείς δεν έχουμε αντίρρηση ε, ε, ε, στο πρασίνισμα, αλλά όντως η γεωργία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Όσον αφορά τώρα το βαθμό πρασινίσματος, είναι κάτι που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ο στόχος θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Πρέπει, να απλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς, να λάβουμε υπόψη τις τοπικές συνθήκες περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, να εξετάσουμε διάφορες από τις υπόλοιπες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μένουν περισσότεροι πόροι εντός της χώρας και όχι να αφαιρούνται. Όσον αφορά το, τον τερματισμό της ειδικής φορολογίας Πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί ούτε σε τοπικό ούτε σε γενικότερο επίπεδο διότι η γεωργία είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να κάνει περισσότερες προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του χρόνου. Τέλος, ε, η Ουγγαρία θέλει να συνεργαστεί επικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τη βάση για τη μελλοντική πολιτική. Ευχαριστώ. Και τώρα ο εκπρόσωπος της Ολλανδικής κυβερνήσεως για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σχολιάσω κατευθείαν αυτό που μας ενδιαφέρει. Η προτάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαπραγματευτική βάση. Όμως θα πρέπει να γίνουν πιο δίκαιε, πιο ευέλικτε και πιο απλέ. Ε, είμαστε υπέρ της ε, δίκαιης ανακατανομής κατανομής ε, των ε, άμεσων ενισχύσεων. Όμως υπάρχει το θέμα της αναλογικότητας και γι' αυτό το λόγο οι προτάσεις που έχει υποβάλει η Κομισιόν δεν είναι αποδεκτές αυτή τη στιγμή. Ή θα εγκρίνουμε ένα ίδιο ποσοστό για, για κάθε κράτος μέλος ή θα μιλάμε για το 4%. Ε, η ευελιξία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη, το είπαν όλοι. Οι προτάσεις Κομισιόν θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτε. Είμαστε υπέρ της προτάσεως του 30% που έκανε η Κομισιόν, όμως να λαμβάνεται υπόψη και η ποικιλία των καταστάσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Ιρλανδός συνάδελφο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση σε κάθε χώρα. Και ασφαλώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την, ε, τον την οικολογική πτυχή, αλλά και άλλα καινοτόμα, και άλλες, και, άλλες, και άλλες καινοτόμες πρακτικές. Είμαστε, μας βρίσκουν σύμφωνοι πολλές από τις προτάσεις που ακούσαμε σήμερα. Ιδιαίτερο συμφωνούμε με, αυτό που είπε, με αυτά που είπε η Γερμανία και η Ιρλανδία σε ό,τι αφορά τους νέους γεωργούς. Και θα πρέπει να βγάλουμε τα κατάλληλα πράγματα από τις, παρου... από τις παλιότερες κρίσεις. Ευχαριστώ. Η εκπρόσωπος της Σουηδίας, κυρία Ντάναν. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία της Υπουργού μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να εκπροσωπήσω σωστά τη χώρα μου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Μας επιτρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα είμαστε επικοδομητικοί. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία εκπρόσωπος της κυβέρνησης της ε, Σλοβενίας, Σιμώνα Μπρέβεκ. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος ε, του Υπουργού μου για την οργάνωση αυτής της συνάντησης. Όλοι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε σημαντικότερα θέματα, τα σημαντικότερα και για μας. Να υπάρχει ευελιξία ε, ως προς τη σύγκληση στα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη διαφέρουν ε, και εάν δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες τους, ε, τότε οι επιπτώσεις είναι βαρισίμαντες. Εμείς χρειαζόμαστε την ευελιξία στη Σλοβενία και είμαστε υπέρ μιας ε, προσέγγισης σύμφωνα με την οποία ε, υπερέχει ο ρεαλισμός. Κατά τα άλλα, προτείνουμε την, ε, στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν, μας μοιάζει διαφανής και καλή και συμφωνούμε και με τη Γερμανία. Η τελική συμφωνία για το τελικό ποσό το τελικό ύψος των κονδυλίων για τις ε, άμεσες ενισχύσεις. Αυτό το πλαφόν ε, θα οριστεί μαζί με τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Εμείς επιθυμούμε να συνεχίσουμε τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές, τη δουλειά που έχουμε ήδη ξεκινήσει στον ε, τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας ε, και θέλουμε να συνεχίσουμε και τη δουλειά που έχουμε αρχίσει στον τομέα της ανάπτυξης της υπέτρου. Συμφωνούμε και με την Αυστρία. Η, η πρόοδος που έχει ε, σημειωθεί μέχρι σήμερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων που έλαβαν το λόγο και προφανώς και όλους τους υπουργούς. Ε, τώρα ε, έχουν απομείνει απλώς κάποιοι βουλευτές που έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν. Κανιέτα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομη ε, σχετικά με την κατάσταση στην Λετωνία και για, θέλω να αναφερθώ στην ε, ε, άνηση μεταχείριση. Περιμένουμε πολλά από αυτή την μεταρρύθμιση και ελπίζουμε να δημιουργηθεί μία, ένας δίκαιος ανταγωνισμός στην Ευρώπη κατά τρόπον ώστε η κοινή αγορά στην Ευρώπη να μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα και να υπάρχουν σωστά κριτήρια όχι όπως στην τωρινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης θεωρούμε ότι η μεταβατική περίοδος πρέπει να είναι πολύ σύντομη, το πολύ τέσσερα χρόνια διότι οι χώρες ε, οι οποίες παίρνουν λιγότερο από το 50% είναι 6 και αυτές ε, πρέπει ε, ήδη να ολοκληρώσουν τη μεταβατική περίοδο και όχι σε 6 χρόνια ή σε 4 χρόνια διότι 30 χρόνια μετά την κατάρρευση του σιδηρού περαπετάσματος γιατί οι χώρες αυτές να λαμβάνουν κάτι παραπάνω από το 50% της μέσης τιμής ακόμη και αν το κόστος παραγωγής διαφέρει, δεν διαφέρει ε, το τριπλάσιο ή τετραπλάσιο και πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε ε, μία λύση ε, μέσω των αμέσων πληρωμών, διότι διαφορετικά αυτό εμποδίζει την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας ορισμένων χωρών. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την α, μεταρρύθμιση πρέπει να πω ότι δεν βλέπω να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές άρα ο προϋπολογισμός δεν αρκεί για τα ε, καθήκοντα τα οποία απαιτούμε από τους γεωργούς. Το έχω πει πολλές φορές και στον Επίτροπο Λεβαντόσχη και στην Επιτροπή, διότι βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και κερδοσκοπία και το ίδιο έγινε με τις χρηματαγορές. Γι' αυτό και εισάγαμε διάφορα μέσα για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή, αλλά στη Γεωργία απομακρυνόμαστε από την παρέμβαση η οποία πρέπει να υπάρχει για τα δημητριακά και σε ορισμένα γαλακτοκομικά διότι θα επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε το εισόδημα και την κατάσταση εις, της αγορές τροφίμων. Θα πρέπει η συνοχή να επεκταθεί στην Ήπερθρο και να υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά το αναγκαίο επίπεδο συνοχής που χρειάζεται. Τέλος πάντων όσον αφορά το πρασίνισμα συμφωνούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι και αυτό είναι πολύ εύκολο όσον αφορά την δημοσιονομική πτυχή. Γι' αυτό και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για την δωρεά διανομή τροφίμων διότι αυτό που κάνουμε δεν γίνεται κατανοητό από την κοινωνία και πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό των τελευταίων 50 ετών της ε, ΚΑΠ για να δούμε τι θα γίνει. Ε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, οι προτάσεις αυτές ε, έχουν καλές αρχές και καλούς στόχους. Αλλά όταν συζητάμε αυτές τις προτάσεις με τους παραγωγούς μας, ε, ακούμε από αυτούς πολύ ανησυχητικά πράγματα. Αυτή η νέα αγροτική πολιτική τι απαντήσεις δίνει έτσι ώστε οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα του ανταγωνισμού ε, που δημιουργεί το, η συμφωνία του Μερκοσούρ για παράδειγμα. Τι απαντήσεις δίνει σε αυτούς τους γεωργούς που έχουν δημιουργήσει μια τεράστια γεωργική κληρονομιά που όμως βλέπουν τις ποσοστώσεις να μειώνονται ή να καταργούνται και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα δεδομένου τη δεδομένης απελευθέρωση των αγορών που υποτίθεται θα αυτορυθμίζονταν. Μήπως θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε αυτές τις προτάσεις. Ποιες είναι οι αποτελεσματικές απαντήσεις που δίδονται έτσι ώστε οι γεωργοί να έχουν ένα σημαντικό κομμάτι από τα κέρδη τα οποία ε, ε δρέπουν άλλοι από το δικό τους υδρότα. Οι διανεμητές ε, και οι μεταποιητές συγκεκριμένα. Τι απαντήσεις λοιπόν δίνει αυτή η καινούργια ε, πολιτική. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ γρήγορα σας παρακαλώ να μιλάτε γιατί βεβαίως πρέπει να δώσουμε το λόγο για να κλείσει ο κύριος Επίτροπος Ράτς Γκαρσία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την οδορία σας. Το πιο σημαντικό αυτή τη μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμα λεχθεί, που είναι ο προπολογισμό. Τι θα γίνει με αυτόν τον προπολογισμό, που ίσω θα είναι ανεπαρκή. Ήδη λέγεται ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε στο 1% του ΑΕΠ. Με το 1% του ΑΕΠ δεν καλύπτουμε ούτε τη σημερινή αγροτική πολιτική. Πολύ δε περισσότερο, πολύ δε περισσότερο τη μελλοντική και με τα νέα κράτη-μέλη. Επίσης, δεν μιλήσαμε για το τι θα γίνει με τις ποσοστώσεις του ζάχαρης. Μετά τη μεταρρύθμιση του 2007, με την τρομακτική προσπάθεια που έκαναν χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, βλέπουμε μια άγρια απελευθέρωση, η οποία υποσκάπτει την βιωσιμότητα του τομέα του κλάδου σε πολλά κράτη-μέλη. Η απελευθέρωση επίσης των δικαιωμάτων φύτευσης Κανένα μέλο του Συμβουλίου δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Η Κομισιόν επιμένει στην απελευθέρωση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα λοιπόν, αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξή. Με αυτή την κοινή αγροτική πολιτική δεν μα εξασφαλίζεται η επιβίωση των επόμενων γενιών, ούτε και η επαρκή ε, προμήθεια τροφίμων τα επόμενα δέκα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να τη σκεφτούμε πολύ καλά αυτή την πρόταση του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα βιοκαύσιμα για τα βιοκαύσιμα ευθύνεται η αύξηση ε, των τιμών των τροφίμων. Αυτό το λένε πάρα πολύ. Πρέπει να προσθέσουμε λοιπόν και αυτό το 3% ε, της καλλιεργούμενης έκτασης. Ε. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε αυτή την πρόταση αν δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα θα δαπανηθούν για τον δεύτερο πυλώνα και πώς αυτά θα καταναμηθούν σε διάφορα κράτη-μέλη. Όμως θέλω να πω το να προσπαθούμε να εξορροπήσουμε ε, τις ε, ε, πληρωμές στα κράτη-μέλη, αυτό πρέπει να είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της ΚΑΠ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες επιμερισμού στο δεύτερο πυλώνα. Ε, και αυτά με βάση ε, διαφορετική μέθοδο ήδη από το 2005. Η πρόταση αυτή καθιστά ε, αντίθετη και ανεφάρμοστη την απλούστευση της όλης διαδικασίας. Στο σύστημα SAPS οι πληρωμές ε, συνδυάζονται με ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε ορισμένους τομείς ε, και δεν ε, αφορά αυτό την ιστορική και παραδοσιακή αξία. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ουγγρικά θέλω να είμαι πιο επιθετική από ότι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ουγγαρίας ο οποίος μίλησε προηγουμένως δεν συμφωνώ με την ανταγωνιστικότητα γιατί για τους Ούγγρους ε, ε, γεωργούς δεν υπάρχει ισότης στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. Οι Πολωνοί και οι Υπουργοί της Πολωνίας εξανέστησαν από τη στάση ε, των γεωργών των πρώην ε, ε, Σοβιετικών Δημοκρατιών και εγώ εξανίσταμαι διότι ελέγχθη ότι μέχρι το 2013 η γεωργοί δεν θα έχουν το ίδιο επίπεδο επιδοτήσεων όσο τα παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές μας στη διακίνηση τροφίμων. Δεν ήταν όμως το, κάτι το οποίο διήρκησε μόνο μέχρι το, που θα διαρκέσει μόνο μέχρι το 2013, διότι δεν νομίζω ότι κανείς επιθυμεί να λύσει το θέμα αυτό. Είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως. Μετά λοιπόν το 2014 αυτή η ανισότητα θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι είναι προδοσία να μιλάμε για τα αγωνιστικότητα διότι ε, όπως και η πολίτες άλλων χωρών όπου υπάρχει λανθασμένη αντιμετώπιση ε, θα υπάρξει ε, σύγκριση και θα προβούν στις ε, σωστές, στα σωστά συμπεράσματα και εάν δουν ότι μειονεκτούν θα εγκαταλείψουν αυτούς τους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ε, αλλά επρόκειτο να ακούσουμε τις απαντήσεις πριν από τις 6.30 τώρα όμως δεν θα προλάβω θα πρέπει να ακούσω τις απαντήσεις στο web streaming στο διαδίκτυο μαζί με όλους τους ανικανοποίητους γεωργούς ανά την Ευρώπη Τώρα θα δοθεί ένα τμήμα των απαντήσεων και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να δώσω το λόγο ε, στον αρμόδιο επίτροπο για θέματα γεωργίας. Τον ευχαριστώ πολύ που ήρθε σήμερα. Για άλλη μια φορά έδειξε ότι είναι πάντα διαθέσιμος να ακούει τις απόψεις και των κυβερνήσεων ε, ε, και των κυβερνήσεων και των ευρωβουλευτών. Και μετά θα μιλήσει ο Μάρσο Τζίτσικη και μετά και εγώ. Κυρία Μορβάη, όταν ανήκουμε σε μια μεγάλη οικογένεια και έχουμε να μοιραστούμε ένα γλυκό, μερικές φορές ε, τίθεται το θέμα το πώς θα το μοιραστούμε. Ο καθένας ε, σκέφτο θα μπορούσε να πάρει ένα κομμάτι μεγαλύτερο από το διπλανό του. Όμως το γεγονός ότι είμαστε όλοι από την ίδια στέγη, ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, ε, μας ε, κάνει να αναρωτηθούμε ε, μήπως είναι καλύτερα έτσι, ε, παρόλο που έχουμε να μοιραστούμε ένα γλυκό και δεν ξέρουμε πώς να το μοιραστούμε, παρά να είμαστε έξω από αυτή την κοινή στέγη. Σας το λέω αυτό καταλαβαίνοντας πολύ καλά βέβαια την απογοήτευση του ενός του άλλου. Όμως έτσι γίνεται κάθε φορά που έχουμε ένα πόρο που είναι περιορισμένος, ένα αγαθό που είναι περιορισμένο και είμαστε μια πολύ τεχνικογένεια. Ωραία. Ως γενική διαπίστωση. Τι βγάζω, τι συμπέρασμα βγάζω από τη σημερινή συζήτηση. Ούτε από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, ούτε από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου δεν άκουσα μια ουσιαστική αμφισβήτηση των στόχων της μεταρρύθμισης ή των βασικών εργαλείων που προτείνονται. Ε, άκουσα σχόλια για το περιεχόμενο αυτών που προτείνουμε, το περιεχόμενο των εργαλείων. Αλλά για το σύστημα των άμεσων πληρωμών, για, το, για τις ε, πληρωμές που θα πρέπει να, είναι, να υποστηρίζουν το βασικό εισόδημα. Ε, πληρωμή για το πρασίνισμα. Τα μέτρα των αγορών στο δεύτερο πυλώνα. Όλα αυτά, για όλα αυτά δεν άκουσα πραγματική απόρριψη. Άκουσα παρατηρήσεις βελτίωσης, βελτιωτικές. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεδομένου ότι είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας διαλόγου. Νομίζω ότι οι προτάσεις μας είναι μια καλή βάση συζήτησης. Είναι συνεπής μεταξύ τους και τα σχόλιά σας είναι συνεπή με αυτά που προτείνουμε. Τώρα, αν πάρουμε τις άμεσες πληρωμές. Έγινε λόγος για τα κριτήρια κατανομής των άμεσων ενισχύσεων. Υπάρχουν δύο απόψει. Αφενός ανάγκη να λάβουμε υπόψη τις, ιδιο... τις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να δώσουμε μεγαλύτερες ενισχύσεις σε συγκεκριμένες ομάδες γεωργών από τις, από τις άλλες. Και από την άλλη μεριά έχουμε την, το στρατόπεδο, ε, την φιλοσοφία ότι θα πρέπει όλοι οι γεωργοί να παίζουν με τους ίδιους κανόνες. Συνεπώς υπάρχει βέβαια το θέμα της δικαιοσύνης και της ισότητας και από την άλλη μεριά υπάρχει το, η ανάγκη να ε, ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα συγκεκριμένων γεωργών σε συγκεκριμένε περιοχές. Πιστεύω ότι με τις προτάσεις μας λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα δύο, γιατί αφενός καταργούμε τις ιστορικές αναφορέ και προτείνουμε κάτι που είναι μετρήσιμο παντού, που είναι οι επιφάνειες που παράγουν τρόφιμα και ταυτόχρονα ε, αποτελούν και δημόσιο αγαθό. Αλλά τις μεταχειριζόμαστε αυτές τις επιφάνειες με διαφορετικό τρόπο. Γιατί δίνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να οριοθετούν περιοχές ε, στις οποίες θα εφαρμόζεται η ενιαία ενίσχυση. Για παράδειγμα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Αυστρία, οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ή μία ε, μόνο περιφέρεια σε όλη τη χώρα, δηλαδή όλη η χώρα να ισοδυνεί με μια περιφέρεια ή να καθορίσει στο εσωτερικό της χώρας διαφορετικές περιοχές, ζώνες για τις οποίες θα ακολουθείται ένα διαφορετικό σύστημα, ένα διαφορετικό ύψος πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις ζώνες. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτό που λέγεται, λέγονται στον τύπο στην Ιταλία, παράδειγμα, ότι ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στο βορρά και το νότο. Όχι, το αντίθετο. Διαβάστε το κείμενο και όταν το διαβάστε θα δείτε ότι έχουμε συμπεριλάβει αυτή την ευελιξία. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και συνέπεια. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και διαφορετικά επίπεδα πληρωμών. Όπως έλεγε και η Σαμπίνα Λαρουέλ, ε, ε, ε, σαν λαζάνια, πράγματι. Σας τρώσαμε λαζάνια. Γιατί, γιατί έτσι είναι και η γεωργία μας. Έχουμε ορεινές περιοχές και παιδινές περιοχές, έχουμε εντατική και εκτατική καλλιέργεια, έχουμε μικρούς και μεγάλους παραγωγούς. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε διαφορετικά επίπεδα και στρώματα. Έτσι, μία διαστρωμάτωση. Ε, όμως, θέλουμε να είμαστε διαφανείς. Τι σημαίνει διαφάνεια για μένα. Να μπορούμε να αποδείξουμε και να δείξουμε πού πάνε τα χρήματα γιατί και να δικαιολογήσουμε γιατί δίνουμε περισσότερα ή λιγότερα στον Α ή το Β. Υπάρχει θέμα ισότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ορισμένοι λένε ότι υπάρχει απουσία πολιτικής βούληση, Ίσως, ίσως. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι την απόφαση θα την λάβουν 27 κράτη-μέλη. Και τα 27 μαζί. Όμω δεν είναι μόνο θέμα πολιτική βούληση, Είναι και θέμα δημοσιονομικών περιορισμών. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω το γεγονό ότι υπάρχει μια χώρα που ε, κάποια χώρα θα εισπράττει πάντοτε τρεις φορές λιγότερα από ό,τι μια άλλη. Κοιτάξτε ταυτόχρονα ποιο είναι το ποσοστό των γεωρικών ενισχύσεων, ε, ποιος είναι το, το, το, ύψος των γεωρικών ενισχύσεων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ Τη κάθε χώρα. Κοιτάξτε και αυτό το κριτήριο. Δεν είναι λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μόνο απόλυτα νούμερα. Ο προπολογισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έλεγε και ο Τζοβάνι Νταβία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι δύο πτυχέ. Για να εξασφαλίσουμε πολιτική απόφαση τελικά. Θα πρέπει να ε, επιταχύνουμε το βήμα μας πολιτικά, σε πολιτικό χρόνο, έτσι ώστε να λυθεί απόφαση πριν το τέλος του 2013. Το σημαντικό δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και το timing. Γιατί αν αργήσουμε πολύ την απόφαση και οι γεωργοί δεν έχουν σαφή νομική βάση το 2014-2015, δεν ξέρω αν το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Τώρα, για το θέμα του πρασινίσματος. Και εδώ τίθεται το θέμα της απλοποίησης και των ίσων όρων. Και εδώ θα πρέπει να ε, έχουμε ε, ευελιξία και στις προτάσεις μας το έχουμε προσπαθήσει. Προσπαθούμε να αναλάβουμε υπόψη ότι οι γεωργοί δραστηριοποιούν σε μία ενιαία αγορά και θα θέλουν αποτελέσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα μέτρα όμως είναι συμπληρωματικά των μέτρων του δεύτερου πυλώνα. Δηλαδή στο δεύτερο πυλώνα μπορούμε να πάρουμε και άλλα μέτρα. Ε, όλες οι προσπάθειες που θα κάνουν οι γεωργοί ε, μέσω των συμβάσεών τους θα, ε, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα θα ληφθούν υπόψη και στον πρώτο πυλώνα. Δηλαδή, ε, στον πρώτο πυλώνα θα πληρωθεί ενίσχυση ε, με βάση τα μέτρα που θα λάβει ε, για να φυτέψει δέντρα. Αυτή η ενίσχυση θα ληφθεί υπόψη στο 7% του δεύτερου πυλώνα. Δεν μιλάμε όμως για γρανάπαυση στο δεύτερο πυλώνα. Ποτέ δεν μιλήσαμε για γρανάπαυση. Δεν είπαμε αφαίρεση, απόσυρση γεών. Μιλήσαμε για οικολογική διαχείριση των γεών. Γιατί, λέω, πολλοί λένε ότι γίνεται ε, ε, ε υπερβολική χρήση ζωοτροφών. Ε, αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Σπατάλη ζωοτροφής. με το 7% προσπαθούμε να έλξουμε γέες που δεν καλλιεργούνται για παράδειγμα σήμερα, βρίσκονται σε αγρανάβαυση και να τις ε, ε, διαχειριστούν οι γεωργοί ε, οικολογικά. Ε, μετά, χρονοδιάγραμμα και προπολογισμό. Η Κομισιόν έχει αναλάβει τι ευθύνε τη. Έκανε πρόταση για τον προπολογισμό. Και θα ήθελα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διατηρήσουν τουλάχιστον το νούμερο που έχουμε προτείνει η νομοθετική πρόταση που έκανε η Κομισιόν έλαβε υπόψη είναι αυτά που πάντοτε προτείναμε για τον προπολογισμό. Τώρα, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα πρέπει όμως να βρούμε μια λύση έτσι ώστε να μην υποσκάψουμε τη δυνατότητα των γεωργών να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της ΚΑΠ. Δεν είναι δυνατόν η απουσία απόφαση για τον προπολογισμό να μπλοκάρει όλα τα υπόλοιπα. Έχετε την υποστήριξή μα έτσι ώστε να πάρετε απόφαση το συντομότερο δυνατόν για τον προπολογισμό. Και το ίδιο βέβαια και για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Για τα μέτρα της αγορά, των αγορών. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την θέση του γεωργού στην αγορά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε υποβάλει προτάσεις. Πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις των αγορών. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει η Κομισιόν να είναι πιο ε, αποτελεσματική αντιδράση Απ' την άλλη μεριά, αν θέλετε να γίνει αυτό, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί η εξουσία τη Κομισιόν. Πώ είναι δυνατόν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε η Κομισιόν να δρά γρήγορα ή να περνάμε από μια διαδικασία η οποία ενδεχομένω θα απαιτεί μήνε για να καταλήξουμε σε μια απόφαση που ήταν ε, ενδεχομένω ορατή εκ των προτέρων. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ποσοστώσεων στου διάφορου τομεί. Ε, το Κοινοβούλιο θα λάβει την έκθεσή μας, πολύ σύντομα την έκθεσή μας για τον τομέα των προεκυπευτικών και θα την εξετάσει. Ε, θα υποβάλουμε έκθεση και για τον τομέα του ίνου. Ήδη ε, έχουμε καταθέσει νομοθετικό πακέτο για το γάλα και τα γαλακτοκομικά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε επίσης την αναδιάρθρωση του τομέα του ελαιολάδου. Συνεπώς όλα αυτά είναι τομεακά ζητήματα και κάνουμε προτάσεις. Υπάρχουν τέτοιοι τομείς και για αυτούς τους τομείς θα υποβάλουμε προτάσεις ή έχουμε υποβάλει ήδη. Μετά, η εχουμε υποβαλει μετα η δίνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να ε, ε, να ε, προσαρμόσουν τις προτάσεις μας μέσω της αρχής της επικουρικότητας. Όμως η αγροτική πολιτική είναι κοινή αγροτική πολιτική. Συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλίζουμε και τη σωστή χρήση των πόρων και των ενισχύσεων. για αυτό το λόγο, όταν μιλούμε για απλοποίηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Μέχρι πού θα φτάσουμε στην απλοποίηση, έτσι ώστε να μην χάσουμε τη δυνατότητα να δικαιολογούμε και να αποδεικνύουμε τη σωστή χρήση των ποσών, των πόρων μας. Τέλος να πω ότι ε, καταλαβαίνουμε την ανάγκη συμβασμού. Θα πρέπει να είναι ένα συμβασμός τελικά πολιτικό ε, που να μην αμφισβητεί τους στόχους μας γιατί αλλιώ θα έχουμε πρόβλημα αξιοπιστία. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική πολιτική που θα είναι ευέλικτη, απλή, αλλά και ταυτόχρονα θα δίνει και αποτελέσματα. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Προσωπικά να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα της συζήτησης, γιατί παρόλες τις ε, αντιρρήσεις που ακούστηκαν, Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο, στην, στο δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. <clears throat> Νομίζω ότι όλοι έχουμε αίσθημα ευθύνης και κατόπιν τούτου είναι φυσιολογικό ότι η ΠΑΚ την οποία θέλουμε να χαράξουμε πρέπει να δώσει και τις σωστές απαντήσεις στους γεωργούς. Πολύ σωστά λοιπόν θελήσαμε να προβάλλουμε αυτή την συνάντηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θέλετε να λάβετε το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι. Και κατόπιν ο κύριος Μάρεξ Σαβίνσκι θα ολοκληρώσει. Μικρόφωνο παρακαλώ, είναι κλειστό το μικρόφωνο του μιλητή. Ναι, λυπούμε κύριε Πρόεδρε που αναγκάζομαι να ξαναπάνω τον λόγο, αλλά χρωστώ μια αναπάντηση στον κύριο Τζον Στουαρτ Άκνιου, ο οποίο ελπίζω να φορεί τα ακουστικά του. Put on your... Yes. θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Άκνιου, κοιτώντα το στα μάτια όπως ζήτησε, ότι η Κύπρος θα αποδεχθεί την πρόκληση για να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσπαθήσει η Προεδρία αυτή να είναι πετυχημένη. Δήλωσε ο κύριος Άκνιου ότι η Γεωργία στην Κύπρο δεν είναι αναπτυγμένη, διότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί είδε μόνο δύο τράκτορς. Φαίνεται ότι ο κύριος Άκνιου επισκέφτηκε τις παραλιακές μας περιοχές και τις τουριστικές περιοχές Ευχαρίστω την επόμενη φορά να το ξαναγήσω και στις γεωργικές μας περιοχές. Ευχαριστώ. Grazie. E adesso... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάρεκ, έχεις εσύ το λόγο για να ολοκληρώσεις αυτή την τόσο σημαντική ημερίδα. Έχουμε ξεπεράσει κατά μισή ώρα το χρόνο μας, αλλά νομίζω ότι μπορέσαμε να δώσουμε σαφείς πληροφορίες και να γίνει κατανοητό ότι οι θεσμοί ε, τους οποίους εκπροσωπούμε επιθυμούν να βοηθήσουν τη Γεωργία. Ο Μάρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας το οποίο είναι αναγκαίο για τη Γεωργία. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε στη συζήτηση αυτή και ιδίως ευχαριστώ τους συναδέλφους υπουργούς και όσοι απουσιάζουν. Φαντάζομαι ότι είχαν κάτι πολύ σοβαρό στις χώρες τους και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο απουσίασαν. Θα ήθελα να τονίσω ότι στη συζήτηση αυτή δεν υπήρχε μόνο δεν υπήρξε ούτε ένας ο οποίος να πει ότι δεν χρειάζεται η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατόπιν 50 χρόνια εμπειρίας και αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, πιστεύω ότι μέχρι στιγμής ακούσαμε διαφορετικές απόψεις ορισμένοι είπαν ότι χρειάζεται μία εκβάθρον αναμόρφωση της κοινή γεωργικής πολιτικής και άλλοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουμε την γεωργική πολιτική αλλά να μην αλλάξουμε τίποτα. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι ένα βασικό στοιχείο αυτού του θέματος είναι ο προϋπολογισμός και τα χρήματα. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση η οποία να επαρκεί για την ευρωπαϊκή γεωργία και ό,τι πόρους έχουμε θα μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, πιστεύω. Θέλω επίσης να τονίσω ότι αναμένω να υπάρξει μία μεταρρύθμιση που θα ορθολογήσει τα θέματα, που θα βοηθήσει τη γεωργία να στραφεί προς το μέλλον. Δεν μπορώ να μιλήσω για τη δικιά μου χώρα, αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να μιλήσω εν ονόματι της Προεδρίας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι μια υποχρέωση η οποία επευλήθη όλους μας και εφόσον υπάρχει μία κοινή γεωργική πολιτική και εφόσον έχουμε, ανα, ε, έχουμε αναθέσει και επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στους γεωργούς για να επιτελούν δημόσιο έργο θα πρέπει όλοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Το πρασίνισμα είναι νέες δημόσιες υποχρεώσεις και στο πρασίνισμα αναφέρεται σε όλους τους γεωργούς ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία προέρχονται. Είναι στον πρώτο πυλώνα και γι' αυτό έχουμε αποδώσει 30% των εθνικών φακέλων σε αυτό το θέμα. 30% Έχουμε λοιπόν πρασίνισμα ή στην Λετωνία όπου θα υπάρχουν λίγα χρήματα μόνο ενώ ή στην Μολδαβία μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότερα. Προσέξτε λοιπόν, δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα αυτό σαν πολιτική τότε ας μην εκπλαγούμε αν μετά από αυτή τη μεταρρύθμιση ακουστούν πολλά παράπονα και υποβληθούν πολλές αγωγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλούμενη διακρίσεις εις βάρος ολισμένων κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ όλους σας, κυρίως τους εισηγητές, οι οποίοι ε, συμμετείχαν σε αυτή την μακρά συνεδρίαση και τώρα καλή τύχη σε όλους. Ε, το έχουμε ανάγκη όλοι. Ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε τη δουλειά, να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο. Νομίζω σήμερα είχαμε μια πολύ καλή μέρα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, αλλά και της αποφασιστικότητας να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός στη σωστή κατεύθυνση. Λύεται η συνεδρίαση.